Ο πρόεδρος, νομίζω ότι εξαντλήσαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Και τώρα να σας τα πω στην μητρική μου γλώσσα, τα πρωτογαλλικά. Uh, Καλησπέρα σας, λέει στα πρωτογαλλικά ο πρόεδρος. Εγώ θα προεδρεύσω σήμερα στη συνεδρίασή μας. Και ξεκινάμε όπως είναι φυσικό με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Πριν εγκρίνουμε τη μέση για διάταξη, πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση για το σημείο 5 όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. θα συζητηθεί αύριο μετά το σημείο 14 στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Οπότε δεν θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί, δηλαδή να συζητηθεί πέμπτο, θα είναι το τελευταίο της αυριανής πρωινής συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Έχετε κάποια ένσταση για την έτσι διάταξη. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε, ας αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Το δεύτερο σημείο μας είναι η έγκριση κάποιων πρακτικών. Από τις 11, ε, 12 Ιουλίου, 1 Σεπτεμβρίου και 5 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προτείνετε, κάποια παρατήρηση. Όχι, επομένως ε, ας θεωρήσουμε εγκεκριμένα τα πρακτικά. Άρα, ξεκινάμε τώρα το ουσιαστικό περιεχόμενο της συνεδρίασης και πρόκειται για το εργαστήρι που αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε την έκθεση σχετική με την ισότητα 2014-2015 που είχε λάβει ο κύριος ε, Ερνέστος Ουρτάσον. Και πρόκειται για αυτό το εργαστήριο να έχουμε κάποιες εισηγήσεις. Συγγνώμη αν δεν πω σωστά τα ονόματα, είναι η κυρία Βιργίνια Λάγκμπακ που είναι η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για Ισότητα των Φίλων. Έχουμε την κυρία Φραντσέσκα Μπετίο που είναι καθηγήτρια οικονομικών στην Σιάννα. Ε, επίσης έχουμε την κυρία είναι και Κλίνγκε. Προεδρεύει τη συμβουλευτική ομάδα για την ισότητα των φίλων ε, για το Horizon 2020. Αυτά προκατακτικά. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ερνέστο Πορτάσον για να μας κάνει την παρουσίασή του. Σε ευχαριστώ Ζωάου και εγώ να ευχαριστήσω τις τρεις εισηγήτριες. Πιστεύω ότι σήμερα θα είναι σημαντική η ημέρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα σχετικά με αυτή την εξαμηνία έκθεση για την ισότητα των φίλων. Ήδη έχουν γίνει κάποιε προκαταρτικέ συζητήσει με του σκιώδε εισηγητέ. Να δούμε ποιε θα είναι οι προτεραιότητέ μα. Έχουμε ήδη ένα πρώτο κείμενο, το έχουμε συζητήσει. Και σήμερα όμω θα τα ακούσουμε από αυτέ τι τρει σημαντικέ προσκεκλημένε ε, που θα μας βοηθήσουν για τις ε, τροπολογίες μας. Θα τις συζητήσουμε. Είναι προτεραιότητα αυτή η έκθεση για να δούμε ποιες είναι οι ρίζες της ανισότητας. Να δούμε ε, επίσης τι προξενεί σήμερα την ε, ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να δούμε ποια είναι η κρατική πολιτική, η πολιτική των θεσμικών οργάνων σε σχέση με το θέμα και τι μπορεί να γίνει. Επίσης προσπαθήσαμε στο σχέδιο κειμένου που ήδη ε, έχουμε εξεργαστεί με τη γραμματεία να θίξουμε όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν την ισότητα. Βεβαίω, θα πρέπει πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ισότητα των φίλων, γιατί πολλά από τα δεδομένα με τα οποία δουλέψαμε είναι στοιχεία που μας τα έδωσε το Ίδρυμα και μα βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε εδώ την διευθύντρια του Ιδρύματος, οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του Ιδρύματος για αυτό το κείμενο. Μας βοήθησε Πάρα πολύ. Αλλιώ ήταν τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Οπότε με την ευκαιρία να την ευχαριστήσω και πάλι. Επίση, έχουμε μια καθηγήτρια ε, οικονομικών. Έχουμε και την κυρία Κλίνγκερ που είναι σύμβουλος για το Ρίζον 2020. Θα μας βοηθήσει να δούμε ε, τι γίνεται με κάποιες άλλες διαδικασίες, κάποια άλλα, ε, ε κάποιες άλλες πλατφόρμες που έχουν σχέση με το Horizon 2020. Να δούμε πού υπάρχει ανισότητα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Εδώ να βάλω τελεία προς το παρόν, να ευχαριστήσω τις συγκήτριες εκ των προτέρων για τα όσα θα μας πούν. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Έρνεστ. Ο θα δώσουμε τις κοιτάλεις στις συγκήτριες και ας ξεκινήσουμε με την κυρία Λάγκμπαρ για την παρουσίαση της. Έχετε το λόγο. Έχετε 15 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος, για την εισήγησή σας. Παρακαλώ, σεβαστείτε αυτό το χρονικόριο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά ε, τις διαφάνειες δεν πρόκειται να σχολιάσω κάθε μία λεπτομέρεια, όμως είναι πολύ σημαντικό ότι πέρα από το δίκτυο, ο οποίος ε, προαναφέρθηκε από τον κύριο Ουρτάσουν, υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα τα οποία προσθέσαμε από άλλες έρευνες, ε, τις οποίες κάναμε σε συγκεκριμένα ζητήματα για τις προεδρίες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω το πώς ήταν η κατάσταση το 2015, τότε είχαμε το δεύτερο δίκτυ. Αν δούμε λοιπόν στη μέση το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι η πρόοδος ε, είναι πάρα πολύ ε, αργή. Ε, το σκορ 52 ανέβηκε μόλις από το 51,3 το 2005, το οποίο σημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων είναι ε, Ένα τομέα πάνω στον οποίο μπορούμε να εργαστούμε πολύ ακόμα. Επίσης έχουμε ε, και τις εξελίξεις, ε, οι οποίες έχουμε και κάποιες εξελίξεις, η περιθεροποίηση, η ισότητα μεταξύ των φίλων ως πολιτικός στόχος, καθώς επίσης και είναι και ένας πολύ σημαντικός τομέας πολιτικές. Κάποια κράτη-μέλη έχουν δει αύξηση πολιτικών κινημάτων που προκαλούν τη γενικότερη ανάγκη για πολιτικές ισότητας των φύλων. Επιπρόσθετα βλέπουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης και τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται και επεκτείνονται από την υπερβολική σεξουαλική βία μέχρι ε, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα κορίτσια, καθώς επίσης και την ακρεοποίηση και τον εξτρεμισμό που επίσης ε, αλλάζουν ε, την δημογραφική κατάσταση των ε, αστικών περιοχών της Ευρώπης ε, και επηρεάζουν φυσικά φτωχούς και πλούσιους. Μιλώντας τώρα για το δίκτυ ε, ισότητας των φύλων, εδώ έχουμε τη γενικότερη εικόνα όπως τη βλέπουμε. Η αύξηση ήταν πάρα πολύ περιορισμένη, διότι παρόλο που κάποια κράτη-μέλη ε, είχαν αύξηση, παρόλα αυτά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρξαν και άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη αύξηση. Οι προκλήσεις λοιπόν παραμένουν και τώρα θα ήθελα να προχωρήσω στον βασικό τομέα εργασίας που αφορά τον τομέα που διασφαλίζει και την οικονομική ανεξαρτησία. Και εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι ένα προαπαιτούμενο για την ισότητα των φύλων, την εξάλληψη της φτώχειας, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, κινείται σταθερά προς το στόχο του 70% για την απασχόληση, όμως ε, όσον αφορά τις γυναίκες το ποσοστό είναι πάντοτε χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Και άμα εξετάσουμε την πλήρη απασχόληση που δεν βλέπετε στην κορυφή της ε, διαφάνειας, όμως άμα δείτε εδώ πέρα το πραγματικό χάσμα παραμένει μεγάλο. Αν το συνδυάσουμε λοιπόν με ε, παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, εκεί βλέπουμε ότι το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ζευγάρι με παιδιά, εκεί το χάσμα είναι το μεγαλύτερο, ενώ ε, μονογονεϊκές οικογένειες, εκεί επίσης το χάσμα είναι πολύ μεγάλο. Βλέπουμε λοιπόν τις διάφορες ε, διαστάσεις των ομάδων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μας. Εδώ έχουμε το σύνολο του πληθυσμού κάτω βλέπετε το ε, χάσμα μεταξύ των φύλων το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ένα ζευγάρι με παιδιά έχει τον μεγαλύτερο, αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα. Σαν παράδειγμα έχουμε μια εικόνα από την Γερμανία εφόσον ε, καταρτίζουμε πληροφορίες με βάση τις χόρτες. Αν συγκρίνουμε λοιπόν χωρίς παιδιά, εκεί δεν υπάρχει κανένα χάσμα. Όμως όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο μεγαλώνει και το χάσμα. Οι οικογένειες λοιπόν με τρία περισσότερα παιδιά πραγματικά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ σοβαρό χάσμα. Αλλά και το χάσμα απασχόλησης είναι στο 43 ε, αν εξετάσουμε τη μερική απασχόληση, που επίσης είναι μία από τις παγίδες που πολύ συχνά ευθύνονται για το χάσμα στην αμοιβή και την απώλεια εισοδημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Το 32% των ε, ανδρών και 9% των ε, ανδρών εργάζονται σε μερική αποσχόληση τέσσερις φορές παραπάνω, δηλαδή οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Επίσης το ποσοστό σε ηλικία μεταξύ 20 και 60, ε, εκεί το ποσοστό είναι 4 φορές υψηλότερο από ό,τι τους άντρες. Στη Μάλτα συγκεκριμένα βλέπουμε ότι ε, πολύ λιγότεροι άνδρες εργάζονται μερική απασχόληση σε σχέση με τις γυναίκες. Το χάσμα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο μεταξύ των δύο φύλων. Η απασχόληση, όπως βλέπουμε, δεν είναι πάντοτε ένα μονοπάτι εκτός της ε, φτώχειας, που βγάζει εκτός της φτώχειας, διότι 9% ε, των γυναικών παίρνουν εισόδημα το οποίο είναι χαμηλότερο από το επίπεδο της φτώχειας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι άμα εξετάσουμε το μεταναστευτικό υπόβαθρο, γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν λιγότερες ευκαιρίες και έτσι λοιπόν κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν εξετάσουμε πάλι τις γραμμές, το μεγαλύτερο χάσμα είναι ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, που έχουν τη λιγότερη απασχόληση σε σχέση με τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί στην ε, Μάλτα, όχι στη Μάλτα γενικότερα. Πάνω από 6 εκατομμύρια ή το 17% των ε, γυναικών χαμηλής χατάρτισης ε, και 12 εκατομμύρια άνδρες μεταξύ 20 ε, και 64 ποτέ δεν έχουν ε, απασχοληθεί. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι όσοι έχουν γεννηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ε, χάσμα μεταξύ τους. Το επίπεδο εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό για την αγορά εργασία και τη συμμετοχή σε αυτήν και όπω βλέπετε για του χαμηλά καταρτισμένου η μεγαλύτερη ομάδα ανέργων είναι οι νεότεροι, όμως το μεγαλύτερο χάσμα είναι όσο αυξάνεται η ηλικία, το οποίο δείχνει και την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες. Επίσης βλέπουμε τη δημογραφική κατάσταση που και το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον. Τα χρήματα τώρα θα ήθελα πάλι να επικεντρωθώ ε, λιγάκι στην εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευση. Άμα δούμε του ε, χαμηλά καταρτισμένου, τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, βλέπουμε εκεί του μη ενεργού. Οι γυναίκε είναι η μεγαλύτερη ομάδα με 49% μη ενεργέ ε, που λόγω δικής τους επιλογής ή της πολυπλοκότητας της αγοράς εργασίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Όσον αφορά τα χρήματα τώρα, οι γυναίκες έχουν το υψηλότερο ποσοστό να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας ε, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, η έλλειψη αυτής πολύ συχνά είναι ένα ζήτημα που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όταν ένας από τους γονείς ή, από το ζευγάρι χάνει την εργασία του, τότε ε, ζευγάρια, ιδιαιτέρως ε, αυτά με παιδιά, αντιμετωπίζουν ε, κίνδυνο νομισματικής φτώχειας. 16% των ζευγαριών με παιδιών κινδύνευαν με φτώχεια το 2014. Εάν όμως ο πατέρας έχανε τη δουλειά, άμα κοιτάξουμε στα δεξιά, με το εισόδημα των ανδρών, τότε η οικογένεια θα βασιζόταν μονάχα στο εισόδημα της μητέρας καθώς επίσης και στα επιδόματα. 70% λοιπόν των ζευγαριών με παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, άμα εξετάσουμε τα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χάσμα μεταξύ των νέων οι οποίοι έχουν λιγότερε πιθανότητε να εργαστούν. Το χάσμα μεταξύ των φύλων μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ηλικία λόγω διαφόρων ε, αιτιών όπως αναφέραμε προηγουμένως το οποίο δείχνει λοιπόν ότι ε, το πώς θα εξελιχθεί η ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική για το έργο μας. Τώρα, για το χρόνο βλέπω, γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες φέρουν την περισσότερη ευθύνη ε, ο συνολικός αριθμός ορών ε, την εβδομάδα που ξοδεύουν οι άνδρες ε, στην εργασία τους ξεπερνά τις 30 ώρες, ενώ στις γυναίκες φτάνει τις 50 ώρες. Αν εξετάσουμε τη μερική αποσχόληση βλέπουμε την πράσινη γραμμή και εκεί μπορούμε να δούμε πώς εργάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες ε, και το σύνολο βέβαια, το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες κάνουν διπλοβάρδιες εργαζόμενες σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ένα ακόμα παράδειγμα από την Γερμανία βλέπουμε τέσσερις φορές περισσότερες ε, γυναίκες εργαζόμενες οι οποίες επίσης μαγειρεύουν, κάνουν το νοικοκυριό τουλάχιστον για μία ώρα την ημέρα. Ο μη ενεργός ε, πληθυσμός, ε, το, το, αναλύσαμε αυτό στη Σλοβακία και ε, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν αναζητούν εργασία. Για το 2005 λοιπόν στη Σλοβακία, από το 2005 μέχρι το 2015, ε, οικογένειες γυναίκες οι οποίες δεν εργάζονται για οικογενειακούς λόγους αυξήθηκε από το 28% στο σχεδόν 40% για το 2015 το οποίο δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι όμως η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Γενικότερα, λοιπόν, το 2005 το 29% των γυναικών ηλικία μεταξύ 20 και 64 δεν ήταν ενεργές. Από αυτές το 30%, 30 δεν αναζητούσαν εργασία, διότι φρόντιζαν τα παιδιά τους ή είχαν άλλες ε, υποχρεώσεις. Ε, και ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για άνδρες και γυναίκες συνδέεται με, την, ε, με, τον, με τη συμμετοχή στην κοινωνία. Όλα αυτά παίζουν λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε να έχουν ένα αίσθημα ότι συμμετέχουν. Ιδιαίτερως οι ε, γυναίκες ε, με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν ε, φράγματα στο, σε ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, σε ζητήματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση, την έλλειψη αυτής, γλωσσικά, γλωσσικά προβλήματα, καθώς επίσης και διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, μιλάμε ε, για ε, την ε, πολυδιάστατη αντίληψη που χρειάζεται να έχουμε πάνω σε αυτό και σε όλο τον κύκλο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Μιλάμε για μονοκονικές οικογένειες, μιλάμε για Ρωμά, ε, μιλάμε για ε, γυναίκες μετανάστριες ε, και αυτό το οποίο συζητάμε ιδιαίτερως αυτή τη στιγμή είναι στόχοι με βάση το φύλλο, είναι μία λύση. Οι πολιτικές ισότητες, ισότητας των φύλων αντιμετωπίζονται ως μαλακές και με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν υπόψη τους όλο το φάσμα. θα πρέπει να εξετάσουμε το τι έχει γίνει και όχι τι έχει επιτευχθεί. Για να κλείσουμε λοιπόν το χάσμα απαιτούνται ξεκάθαροι στόχοι για την ισότητα των φύλων ή στόχοι με βάση τα φύλλα στις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα αυτά, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά και όσον το πολιτές ε, ε, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα βελτιώσει το σχεδιασμό για ε, την επόμενη δράση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Αυτός εδώ είναι ο δείκτης, αν θέλετε να τον εξετάσετε αναλυτικότερα μπορείτε να τον βρείτε στο διαδίκτυο και σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, να πάρετε περισσότερες στατιστικές. Εδώ είναι η διευθύνσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο διεξοδική παρουσίαση. Αλλά στην κυρία Φραντσέσκα Φαρτσέσκα-Βαρτίο. Uh, Καλησπέρα. Ως οικονομολόγος το βρίσκω δύσκολο σε 15 λεπτά να πω κάτι το οποίο δεν είναι κοινότοπο για την ισότητα των φύλων. Πάντως έθεσα το στόχο στον εαυτό μου να εντοπίσω κύριες προτεραιότητες Ξέρω θα συζητήσετε την πλήρη έκθεση αύριο. Μου δόθηκε λοιπόν ένας κατάλογος με σημεία και μιας και το φαινόμενο αυτό είναι πολυέστατο, είναι μακροσκελής ο κατάλογος των σημείων. Θα προσπαθήσω λοιπόν να, να εντοπίσω δύο-τρία σημεία κλειδί που δεν πρέπει να ξεχνάμε από οικονομική σκοπιά και θα πρέπει να καθοδηγούν όλες τις πολιτικές. Για να το κάνω λοιπόν αυτό, θα ξεκινήσω από ένα γνωστό συγγραφέα για αυτά τα θέματα. Τι είναι, εξαφανίστηκε. Κάποιο προβληματάκι υπάρχει φαίνεται. Από τη ΣΥΠΑ, Golding. Η κυρία αυτή είναι ιστορικός οικονομικής ιστορίας και οικονομολόγος. Ανέλησε λοιπόν και αξιολόγησε τις αλλαγές που οι Αμερικανίδες υπέστησαν στη ΣΥΠΑ και ξεκίνησε με αυτή την ήσυχη επανάσταση. Ρωτάω λοιπόν εγώ αρχικά μπορούμε να μιλήσουμε για μια ήρεμη επανάσταση στην οικονομία στην Ευρώπη για τι γυναίκε. Χρησιμοποιώντα βέβαια τις κατηγορίε που θέσπισε η Γκόλντιν. Υποερώτημα. Αυτές οι αλλαγές τι επιτός δέχτηκαν από την κρίση ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ. Η κυρία Γκόλντιν λοιπόν διακρίνει δύο φάσεις στην θέση των γυναικών. Μια εξελεκτική και μια πρόσφατη, την οποία απονομάζει επαναστατική. Μέρος, αυτής της επαναστατικής φάσης είναι η πρόοδη στην απασχόληση. Και μέλος, με κομμάτι της επαναστατικής φάσης είναι κάτι άλλο. Και ιδιαίτερα οι ριζοσπαστικές ριζικές αλλαγές σύμφωνα με αυτή την ιστορικό σε τρεις όσον αφορά τι επιλογέ των γυναικών και την ε, λήψη των αποφασιών του. Α δούμε ποιε είναι. Καταρχά, η πρώτη αλλαγή αφορά τον ορίζοντα, όπω λέμε. Διαβάζετε στα μικρά γράμματα, είναι η επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και το κατά πόσο η γυναίκα αποφασίζει να δεσμευτεί πλήρως ή εν μέρη όσον αφορά τον τομέα εργασία. Εντάξει, το δεύτερο και αυτό ενδιαφέρον, αλλά με ενδιαφέρει κυρίω η τρίτη αλλαγή, δηλαδή η διαδικασία λήψη απόφαση. Εδώ, όπως θα διαβάσετε, η διάκριση είναι το κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις οι εργασιακές λαμβάνονται από κοινού, αν μια γυναίκα είναι παντρεμένη βρίσκεται σε μακροχρόνια σχέση ή αν η γυναίκα είναι αυτός ο, δεύτερο δεύτερος εισοδηματίας του σπιτιού και τι γίνεται με τις αποφάσεις που αφορούν την εργασία. Η αντίθεση λοιπόν είναι εδώ μεταξύ απολύτως κοινών αποφάσεων στα πλαίσια του νοικοκυριού σε σχέση με τη θέση ενός δεύτερου συμβάλλοντα σε εισόδημα στο σπίτι και πώς λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις και πώς κάνει τις επιλογές της. Από οικονομική λοιπόν σκοπιά, η λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμη σημασία. Κάνουμε λοιπόν το εξή ω άσκηση. Μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν έχουν, στην Ευρώπη δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα όσον αφορά τις ύπες σχέση με την ταυτότητα και τον ορίζοντα. Έτσι, μιλάω για τα πρώτα κριτήρια θεωρώ δεδομένο ότι ήδη έχουν λάβει χώρα κάποιες αλλαγές και είναι αρκετά έντονες. Τώρα, σε σχέση με την ε, λήψη των αποφάσεων. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζω τρία κρίσιμα κενά. Τα δύο είναι σχετικά γνωστά, το τρίτο λιγότερο. Κοιτάξτε αυτή την γραμμή Διαφορέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια εξέλιξη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με κάποιες αλλαγές και είχαμε κάποια πρόοδο πρόσφατα, αλλά όχι τόσο σημαντική. Τα τελευταία στοιχεία μας δείχνουν ένα έλλειμμα, ένα κενό 16,2. Υπάρχει πρώτο αλλά οι αλλαγέ δεν είναι μεγάλε. Το δεύτερο κενό που θα δείτε και το οποίο μάλλον γνωρίζετε είναι η σύνταξη, το ύψο τη σύνταξη και κατά πόσο ποικίλει από άντρε και γυναίκε. Αυτή είναι η πράσινη γραμμή σε σχέση με τη ΜΟΒ προηγουμένω. Θα δείτε εδώ το κενό αφορά τα στοιχεία τελευταίων ετών είναι 40% και είναι σχετικά σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες κατά μέσο όρο κερδίζουν 40% λιγότερο όσον αφορά τι συντάξει σε σχέση με του άντρε. Και μετά έχουμε τις κόκκινες στιγμές, το άλλο κενό, 40% και πάλι περίπου, και όπως βλέπετε φαίνεται να έχει μειωθεί δραματικά. Τι είναι αυτό το κενό. Αυτό είναι ένα άγνωστο μέχρι τώρα κενό, γνωστό στους στατιστικολόγους κυρίως. Αυτό που ονομάζουμε συνολικό κενό ή διαφορά στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τι σημαίνει, είναι σχετικά απλό. Αν πάρουμε όλους τους άντρες και όλες τις ε, γυναίκες από τα 15 μέχρι τα 64, τι κάνουμε, προσθέτουμε το εισόδημα που φέρνουν οι γυναίκες στο σπίτι, σε αυτές που δουλεύουν, αλλά και αυτές που δεν δουλεύουν. Κάνουμε το ίδιο για τους άντρες, παίρνουμε το μέσο όρο και το διαιρούμε και βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο όλες οι γυναίκες μαζί συμβάλλουν στο νοικοκυριό γύρω στο 40% λιγότερο από ότι οι άντρες. Πολύ κοντά δηλαδή στο κενό που αφορά τις ε, συντάξεις σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Όπως θα δείτε λοιπόν, αυτό το κενό υποχώρησε κατά διάρκεια της κρίσης από το 44% στο 41% και μετά έμεινε σταθερό τα πρώτα χρόνια της κρίσης, έτσι. Και ένας από τους λόγους είναι ότι οι γυναίκες τα κατάφεραν καλύτερα κατά διάρκεια της κρίσης από ότι οι άντρες, κατά κάποιο τρόπο, και υπήρξε μια εξισορρόπηση από κάτω. Οι, γυναίκες, οι άντρες λοιπόν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν τα κατάφεραν τόσο καλά όσο οι γυναίκες, γι' αυτό ακριβώς φαίνεται περισσότερη ισότητα για τις γυναίκες και σταθερότητα. Έχουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο πράγμα για να προοδεύσει λοιπόν κανείς όσον αφορά την ισότητα των φύλων από οικονομική σκοπιά, θα πρέπει, Όπω λέμε στην Αμερικανική αργό, ποιο φέρνει το μπέικον στο σπίτι. Και υπάρχει τεράστια διαφορά εδώ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε τι οφείλεται τώρα. Θα δείτε εδώ ότι η κατανομή αυτού του κενού του 40% ακολουθεί μια κατανομή. Εδώ το μαύρο αφορά το ότι πολύ λιγότερες γυναίκες και μετά άντρες δουλεύουν. Το κίτρινο αφορά την ε, αμοιβή ανά όχι, η αρθένια μιλήτρια. Το κίτρινο οφείλεται στο γεγονό ότι παρόλο που οι γυναίκε εργάζονται, εργάζονται λιγότερε ώρε από του άντρε. Και η πορτοκαλί γραμμή αφορά το γεγονό ότι σε ωραία βάση οι γυναίκε αμείβονται περίπου 16% λιγότερο από ότι οι άντρε. Οπότε βλέπετε ότι τρει αυτέ συνιστώσει αθρίζονται στο 40%, στο ποσό αυτό το 40%. Αυτό που θέλω να τονίσω στο χρόνο που μένει τώρα είναι ότι η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτό το θέμα θέτω και δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό, αλλά πάνω το θέτω το ερώτημα, οι οικονομικές μας πολιτικές που χαράσουμε ως Ένωση, κατά πάσα πιθανότητα με τρόπο επιθετικό θα αντιμετωπίσουν και θα βελτιώσουν αυτό το κενό. Τώρα, εδώ έχουμε δύο ζητήματα που βλέπω έτσι να είναι στη μέση. Το ένα είναι το θέμα της μερικής απασχόλησης που ανέφερε και η Βιρτζίνια. Θα δείτε εδώ λοιπόν σε κάποια στοιχεία ότι μία από τις τόσα στη διαφορά αμοιβή οφείλεται στο γεγονό ότι οι γυναίκες εργάζονται πολύ λιγότερες ώρες. Οπότε το θέμα εδώ της μερικής απασχόλησης δεν έχει τόσο να κάνει. Εντάξει. Και τώρα, πώς πάνε τα πράγματα από αυτή την άποψη. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Μεταξύ 2000 και 2015 η καθαρή αύξηση απασχολησιμότητας στις γυναίκες στις 27 χώρες της Ένωσης, όπως βλέπετε εδώ, ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Στη μερική απασχόληση είχαμε 7 εκατομμύρια. 70 λοιπόν περίπου της 100 της καθαρής αύξησης στην γενική απασχόληση αφορά και οφείλεται κυρίως στην μερική απασχόληση, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 70% λοιπόν. Εντάξει. Και λόγω αυτού του γεγονότος, μία στις τέσσερις γυναίκες σε μερική απασχόληση είναι παρά τη θέλησή της σε μερική απασχόληση, δηλαδή θα ήθελε να δουλεύει περισσότερο. Παρόλο λοιπόν που βελτιώσαμε την απασχόληση για τις γυναίκες, βλέπουμε τον αριθμό των ωρών να μειώνεται. Αν ανατρέξουμε λοιπόν στους στόχους μας, δηλαδή σωστέ αμοιβέ για τι γυναίκε σε σχέση με του άντρε, τότε θα δούμε ότι αυτά τα δύο πάνε σε αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μπορείτε να βελτιώσετε τον δίκτυο απασχόληση, αλλά μειώνετε τι ώρε απασχόληση. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι ένα θεματάκι και το οποίο θα πρέπει να εξισορροπηθεί. Ένα άλλο ζήτημα δεν είναι το εξή. Η Ευρώπη είναι διχασμένη, όπως ξέρετε κι εσείς, οικονομικά έτσι, όχι, δεν μιλάω πολιτικά. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, εδώ το θέμα ποικίλει, εικόνα ποικίλει. Αν κάνετε μια απλή άσκηση, θα σας δώσω λεπτομέρειες αν θέλετε, και πείτε ότι το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ακολουθεί το μέσο όρο βάσης που είχαν παρατηρήσει μεταξύ του 2 και του 12 πριν και μετά την κρίση δηλαδή κατά μέσο όρο. Πόσος καιρός θα χρειαστεί οι γυναίκες να πετύχουν το στόχο του 75% απασχόλησης πλήρους, ε, ολικής, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι και τμήμα της στρατηγική 2020, έτσι. Για την Ευρώπη των 27, λοιπόν, θα χρειαστούν τα χρόνια μέχρι το 2037. 2037 για το σύνολο της Ένωσης. Όμως, αν εξαιρέσουμε τις χώρες όπου η γενική απασχόληση είναι στο χαμηλότερό της και αυτές οι χώρες πολύ συχνά είναι οι χώρες οι οποίε ε, επλήγησαν περισσότερο από τη λιτότητα και την κρίση γενικότερα. χώρες δηλαδή όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, ε, ίσως και άλλες που είπα ξέχασα. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε αυτές τις χώρες, μάλλον αν πάρουμε αυτές τις χώρες και επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία, τότε θα χρειαστεί με το 2062 για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν κρίνουμε την πρόοδο στην ισότητα των φύλων από οικονομικούς όρους στην Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Δηλαδή η πρόοδος θα πρέπει να είναι ταχύτερη και όχι αργότερη στις χώρες οι οποίες υπολείπονται. Και τώρα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο να ισχύει. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Έτσι. Καταλήγοντας λοιπόν, αν συμφωνήσουμε με την άποψη του Κόντιν ότι η πρόοδος στην απασχόληση των γυναικών αποτελεί ένα εξελικτικό προαπαιτούμενο για να γίνουν ριζοσπαστικέ αλλαγέ. Αυτό λέει τουλάχιστον η κυρία Γκόλτινγκ, έτσι. Αυτό λέει τουλάχιστον για Αμερική στη σύνοψή τη. Τότε στην Ευρώπη, στην Ευρώπη θα πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά ακριβώ τα προαπαιτούμενα τα ίδια. Η κρίση που είδαμε εξίσωσε τη θέση των ατόμων στην αγορά εργασία προ τα κάτω υπάρχει περισσότερη ισότητα προς τα κάτω για όλους. Η πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στην Ευρώπη σε επίπεδο ισότητας απέχει πολύ ακόμα από την υλοποίηση, γιατί ακόμα έχουμε ένα 40% απόκληση στις αμοιβέ. Και ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι οι τρονές οικονομικές μας πολιτικές στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο ύψος των περιστάσεων. Εκεί το αφήνω αυτό εκκρεμές σε ερώτημα, γιατί έχω περάσει και 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ίνικε Κλίνκε, η οποία θα κάνει την τελευταία στις παρουσίαση και κατόπιν θα γίνει συζήτηση. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, με καλέσατε και με τιμά η πρόσκλησή σας για να σας μιλήσω σήμερα το απόγευμα για να δούμε τώρα τι γίνεται με τη διάσταση του φύλου. Πώς δηλαδή μπορεί να έχουμε μία ανάλυση ε, των φύλων ούτε ώστε να έχουμε όσον αφορά την καινοτομία αριστεία. Δεν ξέρω πόσο αυτό σχετίζεται με την ε, έκθεση την οποία τώρα συντάσσεται αλλά μου είπαν γι' αυτό να σας πω. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι σαν το χρυσό κανόνα γιατί αφορά τις ε, ανάγκες των γυναικών και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ε, αριστεία στην ε, έρευνα και αυτή η ανάλυση είναι τμήμα της έρευνας σχέση με την αριστεία σε σχέση με την γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία ώστε να έχουμε εμπορεύματα και υπηρεσίες που να είναι πιο βολικά για τις ε, δυνάμει αγορές και να λαμβάνει υπόψη και το θέμα των στερεοτύπων. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται να καταβληθούν κάποιες προσπάθειες ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ένταξη του θέματος των δύο φύλων ε, στους κεντρικούς άξονες πολιτικής. Οπότε θα πρέπει από τη χάραξη πολιτικής να είναι κάτι που κάθε μέρα να μας απασχολεί σε κάθε πρόταση, σε κάθε αξιολόγηση. Αυτό θα να δούμε γιατί το θέμα είναι τόσο κρίσιμο. Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα σε σχέση με το Horizon 2020 και πώς όλα αυτά αντικατοπίζονται στις ε, δραστηριότητες της δικής μας ομάδας, της συμβουλευτικής ομάδας για τα θέματα των δύο φίλων. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις, να δούμε ποιες είναι οι άριστες ε, πρακτικές, τι συστάσεις μπορούμε να κάνουμε τώρα όσον αφορά τους στόχους του ορίζοντα 2020 και τους στόχους για τα δύο ε, φύλλα, ξέρετε τα πράγματα πως έχουν και εγώ θα επικεντρωθώ στον τρίτο στόχο, δηλαδή το τι γίνεται με τα δύο φύλλα όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Για να είμαι πιο ξεκάθαρη, να σας πω ακριβώς τι εννοούμε με αυτή τη διάσταση των δύο φύλων γιατί βασιλεύει σύγκριση. Δεν είναι θέμα συμμετοχής των γυναικών στην λήψη αποφάσεων και στην έρευνα. Δεν είναι θέμα θεσμικών αλλαγών και έτσι να είναι πιο φιλικά τα θεσμικά όργανα, αλλά είναι κάτι που αφορά το περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας και συγκεκριμένα είναι θέμα της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας. Οπότε τελικά πρόκειται για το πώς θα κινητοποιήσουμε νέες μεθόδους και να είναι πιο συνεπείς η επιστημονική υφή αυτών των ερευνών. Έχουμε τώρα κάποιε γνώσεις για το πώς οι διαφορέ των δύο φύλων, οι βιολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν στην βιολογία, την ιατρική, αλλά και αλλού. Να, ας πούμε στα θέματα περιβάλλοντος, μεταφορές, ασφάλεια οχημάτων, ε, διαστημική ιατρική κλπ. Αυτό ίσως είναι κάτι το καινούριο ε, είναι πιο δύσκολο να το εξηγήσουμε, αλλά θα πρέπει κανείς να μην ξεχνάει τα θέματα συμπεριφοράς των μεν και των δε. Πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν έρευνα και καινοτομία και πολλές φορές ε, υποσυνείδητα, συνέστητα και ε, η ανάλυση των διαφορών των δύο φύλων προσπαθεί να το ξεπεράσει. Μα εμείς δεν θέλουμε οι κανόνες που βασίζονται στα στερεότυπα να επηρεάσουν την καινοτομία και την έρευνα. Γιατί αν γίνει αυτό, τότε θα χαθούν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά και πολύ χρήμα. Να, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σταματήσουμε την ενιαία αντιμετώπιση. Θα πρέπει η έρευνα και η τεχνολογία να ανταποκρίνεται πιο υπεύθυνα στις διαφορετικές ανάγκες των δύο φύλων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιους ε, άλλους παράγοντες σε σχέση με ηλικία, εθνοτική προέλευση, σεξουαλικό προσανατολισμό και βέβαια φύλλο. Τώρα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το Horizon 2020 και για την λήψη υπόψη των δύο φύλλων έχουμε ένα project που είναι η δέουσα μέθοδος. Ξέρετε τι είναι η ήδη Έχουμε ένα website, έχουμε και κάποιες δημοσιεύσεις. Ε, και στα πλαίσια του 2020 οι ετούντες παραπέμπονται εκεί, σε αυτό το υλικό, όταν υπάρχει κάτι το οποίο επηρεάζεται από τη σχέση των δύο φύλων. Επίσης ε, έχουμε ε, αναπτύξει και κάποια και studies ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα γνώση, πιο κατάλληλη, πιο ταιριαστή στο κάθε φύλλο. Και αυτό σε όλους τους τομείς του ορίζοντα 2020, βιοιατρική, ε, πειράματα, ε, καρδιοαγγειακά, δημοσία υγεία, ε, καρκίνος, νοοτεχνολογία μη μεταδόσιμες νόσους, ε, επίσης ε, τεχνολογία που βοηθά τους πιο ηλικιωμένους σε όλα αυτά, σε όλα αυτά ε, θα πρέπει αυτός ο παράγοντας να ληφθεί υπόψη και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο website μας. Οπότε για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Είμαστε στο μισό της διαδρομής που οδηγεί στο ορίζον 2020. Έχουμε κάποια θέματα που θεωρούνται προτεραιότητας και αυτοί που συγκρότησαν το πρόγραμμα θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα δύο φύλλα. Έχουμε τη συμβουλευτική ομάδα, εντολή της είναι να παράσχει συμβουλές στην Κομισιόν. Ιδίω όσον αφορά τη λήψη υπόψη της διάστασης των δύο φύλων. Δύο-τρεις φορές το χρόνο συναντώνται και συμβουλεύουν για διάφορα θέματα ε, για το πρόγραμμα εργασιών του 2014-2015, 2016-2017, αλλά και για το επόμενο Οπότε όλα αυτά έχουν βοηθήσει τη στρατηγικό σχεδιασμό με διάφορες ιδέες που φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση με τα δύο φύλλα. Επίσης έχουμε επεξεργαστεί και κάποιες δικές μας πρωτοβουλίες όπως τις κατευθυντήριες για την επιλογή των αξιολογητών που θα έχουν εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα των δύο φύλων και πτήσουμε και άλλες δραστηριότητε φέτος Οπότε για να δούμε ποια είναι τα πλέον επιγόντα σήμερα. Δύο θα σας αναφέρω. Πρώτον, να βελτιώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης για τις προτάσεις όσον αφορά τη διάσταση της όντας των δύο φύλων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η αξιολόγηση γίνεται στα σοβαρά και δεόντως. Ε, επίσης, θα πρέπει να ε, μεγιστοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη των αξιολογητών. Οπότε, για να δούμε τώρα πώς θα είναι καλύτερη η αξιολόγηση των προτάσεων. Οι προτάσεις αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις, την εφαρμογή, την αστεία και στην αριστεία λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και ζυγίζεται. Όμως αυτό το οποίο επιδέχεται βελτίωση είναι το πώς όλα αυτά σε συγκεκριμένα θέματα θα επιληθούν, θα διεκπαιρεωθούν. Γιατί υπάρχει εδώ ένα κενό μεταξύ της πολιτικής και της πρακτικής. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα εκεί που θα πρέπει υποχρεωτικά να βάλουν την υπόψη των δύο σε αξιολόγηση. Επίσης υπάρχει αυτό το κενό και το αποτέλεσμα ποιο είναι ότι δεν εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες της ε, ανάλυσης. Και έτσι πάσχουν και οι επιδόσεις της κάθε προσπάθειας. Αυτό είναι απογοητευτικό. Ιδίω για τους ειδικού οι οποίοι έχουν επισημάνει την πράγμα γίνεται ανάλυση επιβεβαίωσης των των δύο φύλων. Και αυτό σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου γιατί τον Δεκέμβριο του 2015 σημείο 9 θα το Σύμβουλο από την Κομισιόν να λάβει υπόψη τα θέματα των ε, δύο φύλων εν ώψη του ορίζοντα 2020 και στι διαδικασίε αξιολόγηση, πιστεύω. Επίση, θα πρέπει αυτή η διάσταση των δύο φύλων να θεωρηθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την ε, μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και αναδιόριση, Οπότε, να δούμε ποια είναι η προσθεμένη αξία από αυτή την προσπάθεια και για αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει έτσι να οδηγηθούμε σε καλύτερες επιδόσεις για τα αποτελέσματα, για την αξιολόγηση, για όλα. Και το Καναδικό Ίδρυμα Υγείας όλα αυτά τα έχει λάβει υπόψη ε, και τα έχει ποσοτικά αξιολογήσει όσον αφορά τα, θέματα βιοιατρικής έρευνας. Κατά τη γνώμη μου, επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βοηθήσουμε στην συμπερίληψη αυτού του κριτηρίου, τη διάσταση τη ισότητα των δύο φύλων, σε όλα τα προβλήματα. Και βέβαια να δεχθούμε ότι έχουμε και κάποιες θεμητέ εξαιρεσει που βέβαια θα υποστηρίζονται από κατάλληλη επιχειρηματολογία για να χαρακτηριστούν τέτοιες. Τώρα για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η αξιολόγηση to uh, what was the solution to my first problem. The second problem is to... Ε, Άρα, συγγνώμη, σε έλεγα το πρώτο με το δεύτερο. Θα πρέπει να δούμε επομένω πώ θα βελτιώσουμε του αξιολογητέ. Γιατί ζητάμε πάρα πολλά από του ερευνητέ και από του ετούντε. Του έχουμε δώσει τα εργαλεία από το project για την καινοτομία. Αλλά θα πρέπει να καλύψουμε και τι ανάγκε αυτών των αξιολογικών. Πέραν τη σύντομη ε, ενημέρωση πριν κάνουν την αξιολόγηση, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα διότι Κατά κάποιο τρόπο αυτοί αξιολογητέ θα πρέπει να είναι ακόμα πιο καταρτισμένοι όταν κάνουν την αξιολόγηση του σε σχέση με του ετούντε. Άρα χρειάζεται κάποια κατάρτιση, κάποια εκπαίδευση αυτών. Και πάλι στον Καναδά ξέρουμε ότι έχουν κάποια κατάρτιση online, ιντερνετική για όλες τις αιτήσει, ούτως ώστε να αυξηθεί η δεξιότητά τους, η ικανότητά τους στην αξιολόγηση και κατόπιν αυτής της κατάρτισης δίνεται και ένα σχετικό πτυχίο. Επίσης, στις κάτω χώρες τώρα έχουμε ένα νέο ελληνικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται ε, «Φίλο και Υγεία». Ε, έχει υποστηριχθεί με 20 εκατομμύρια από την κυβέρνηση και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ορίζον 2020. Πώς δηλαδή θα δίνονται οδηγίες στους τούντες, αλλά και πώς θα δίνονται οδηγίες στους αξιολογητές. Να, αυτά είναι τα εργαλεία που έχουν. Προσπάθησα όσο μπορούσα να σας τα εξηγήσω. Να, και εγώ βλέπουμε επίσης τι εργαλεία έχουν χρησιμοποιήσει οι Καναδοί για την ε, βιοιατρική έρευνα, ε, για τη δημοσία υγεία και σχετικούς τομείς. Τώρα, να σας πω τις ε, συστάσεις μου εν τέλει. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατανόησή μας της διάστασης της όντως των δύο φύλων. Να μην υπάρχει ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Να μην υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ πρακτικής και στρατηγικής ή πολιτικής. Να μπορούμε να έχουμε απόδοση των επενδύσεων που κάνουμε στα project μας. Να υπάρχει κατάλληλη ανάλυση για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ε, δημιουργικότητα των νέων ερευνητών. Και σας ευχαριστώ. Eh, e Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για τις πολύ καλές ε, παρουσιάσεις τους, ε, καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες ε, που μας έδωσαν. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας, η οποία δυστυχώς όμως θα πρέπει να είναι σύντομη. Όμως ε, μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά ε, στα μέλη, η κυρία Κοβλόφσκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, για ε, τα όσα είπανε. Συγκεκριμένα όσον αφορά την παρουσίαση από την ε, κυρία Φραντσέσκα ε, Μπιέτο, η οποία παρουσίασε το χάσμα ε, δεν μιλάμε πάρα πολύ για αυτό και νομίζω ότι όλα αυτά ε, τα στοιχεία είναι καλοί δείκτες για το επίπεδο ισότητας των φύλων. Αν αναρωτιόμαστε λοιπόν το πού βρισκόμαστε στην ε, καταπολέμηση της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα του χάσματος όσον αφορά τη σύνταξη αλλά και τις αμοιβέ. Οι δείκτες αυτοί όμως είναι μερικοί διότι δείχνουν μονάχα ένα κομμάτι της εικόνας ε, το ολιστικό χάσμα λοιπόν κατά τη γνώμη μου ε, είναι οι καλύτεροι δείκτες ε, που συλλέγουν και δείχνουν όλες τις ανισότητες στις καριέρες των γυναικών. Όταν μιλάμε για το χάσμα στον μισθό αυτό μονάχα αντικατοπτρίζει μονάχα ένα κομμάτι Η θέση της λοιπόν, όλες οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών συλλέγονται και φαίνονται ε, στο ε, συνταξιοδοτικό χάσμα. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό για εμάς να αντιμετωπίσουμε το χάσμα αυτό ως το πιο επίσημο δείκτη και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και θα πρέπει να αναζητήσουμε και ε, μεθόδους ε, για την αξιολόγηση αυτού του χάσματος και με μια ενοποιημένη μέθοδο θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που εφιστήσατε την προσοχή μας σε, αυτά, σε αυτούς τους σημαντικούς δείκτες για τους οποίους δεν συζητούμε παρκώς. Γίνεται λοιπόν κάτι ε, σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου, όχι αρκετά όμως, νομίζω όμως ότι είναι η αρχή από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας ειλικρινής καθρέφτης ο οποίος θα μας δείξει το που βρισκόμαστε ε, για την, στην μάχη για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ε, μεγάλη εντύπωση μου έκανε η διαφάνεια όπου παρουσιάσατε τα μέρη τα οποία επηρεάζουν όλο αυτό το χάσμα. Είναι ενδιαφέρον διότι έχουμε ένα χάσμα στην απασχόληση και σε αυτό προσθέσατε τον αριθμό ροών στη δουλειά καθώς επίσης και άλλες ανισότητες όπως είναι για παράδειγμα ε, η ε, κορυφή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 της τάξης ε, και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να είναι η βάση ε, για τις ε, πολιτικές ισότητας και η βάση για να προετοιμάσουμε εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να αποτρέψουν αυτό το χάσμα στη σύνταξη. Θα υπάρξει μια αναφορά από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα για τα ε, συνταξιοδοτικά συστήματα, όμως δεν είναι αυτά η αίτια πίσω από το πρόβλημα, διότι η σύνταξη που παίρνει είναι η συνέπεια του πώς λειτουργούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Και έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Όλα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ήταν σημαντικά για τη συζήτηση που κάνουμε και για τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και τα οποία έχουν και σημαντικούς αριθμούς. Ε, δύο θέματα όμως με απασχολούν εμένα. Ε, επανειλημμένως αναφέρθηκε, είχαμε μια παρουσίαση, ο ανδρικός πυλώνας και ο γυναικείος πυλώνας ε, δεν είναι ε, πυλώνες οι, οποίοι, πυλώνες οι οποίοι βρίσκονται δίπλα-δίπλα αλλά που επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ποσοστό εισοδήματος των γυναικών βρίσκεται στον νόμο των γυναικών και θα με ενδιέφερε λοιπόν πώς ε, οι σχέσεις αυτές μπορούν να εξεταστούν καλύτερα διότι το θέμα αφορά ότι οι υψηλές δυνατότητες ε, για μία σύνταξη πέφτουν στους ε, ώμους των γυναικών και οι γυναίκες ε, συνεισφέρουν ούτως ώστε οι άνδρες στη συνέχεια να πάρουν μία υψηλότερη σύνταξη. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς αυτούς τους δύο πυλώνες μπορούμε να τους εξαντάσουμε από κοινού και επίσης το ποσοστό απασχόλησης. κατάγουμε από τη Γερμανία και στη Γερμανία πάντοτε μιλούσαμε ώστε να προωθήσουμε την υψηλή απασχολησιμότητα των γυναικών. Διότι σε περίπτωση που καταφέρουμε αυτό, λέγαμε, τότε θα έχουμε πραγματική ισότητα. Όμω, εν τέλει, συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα δύο δεν συσχετίζονται. Οι γυναίκε να απασχολούνται περισσότερο, όμω αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να ζήσουν με τα χρήματα τα οποία βγάζουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν στο μέλλον θα υπάρχει ένα άλλο παράγοντα ή δείκτη στο επίκεντρο σχετικά με το αν μπορούμε να ζήσουμε με τα χρήματα που βγάζουμε, διότι το ότι έχω μία 40ωρη δουλειά δεν λέει απολύτω τίποτα σχετικά με το αν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τα χρήματα που βγάζω. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίες δουλεύουν 40 ε, ώρες την εβδομάδα, όμω ταυτόχρονα φροντίσουν παιδιά και ηλικιωμένους στο σπίτι και ταυτόχρονα δεν μπορούν να τα βγάλουν όλα αυτά, γιατί η απασχόληση είναι τόσο χαμηλή. Έτσι λοιπόν το ερώτημα, εάν αυτός ο παλιός δείκτης σχετικά με την ποσόστοση στην απασχόληση μας ενδιαφέρει ακόμα ή θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα νέο δίκτυο ο οποίος θα ορίζει εάν μπορώ να ζήσω με τα χρήματα που βγάζω ασχέτως με τα πόσες ώρες ε, δουλεύω. Ευχαριστώ κύριε Ανόηλ. Ο κύριος Μέντα Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αμφισβήτητο ότι οι τρεις μας εισηγήτριες μας έδωσαν πλήρες και κέρδιες πληροφορίες για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει πολύ υλικό για το οποίο θα μπορούσαμε να συζητάμε εδώ και στη δική μας Επιτροπή αλλά και σε άλλες Επιτροπές του Κοινοβουλίου. Αυτά που μας είπαν οι συγγήτριες μας αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μία αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενισχύονται όλο και περισσότερο σε κοινωνικό επίπεδο. Και οι ίδιες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξάνονται. Και δεν είναι τυχαίο σήμερα στην Ευρώπη των 28 ότι το 1 τέταρτο αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας. Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε 20 εκατομμύρια άνεργους στο εσωτερικό της Ένωσης. Εδώ μιλάμε λοιπόν για δεδομένα, λεπτομερή και αναλυτικά, τα οποία όμω καμιά φορά να μπορεί και να παρουσιάζουν κάποια στρεπλή εικόνα της απασχόλησης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι υπολογίζονται ως μη ενεργοί στην αγορά εργασία και αυτό όμως συμβαίνει όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Οπότε ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει άμεσα και ίσως θα πρέπει εδώ να κάνουμε και μια πολιτική συζήτηση και ανάλυση, είναι το εξή. Ωραία. Αυτό είναι το σενάριο που έχουμε μπροστά μα. Αλλά αυτό οφείλεται σε κάτι, έτσι. Πού είναι τα αίτια, τα συγκεκριμένα αίτια που αποτελούν την βάση τη επιβάρυνση και τη συνέχισης αυτή τη κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά από ένα σενάριο όπως αυτό που μας παρουσίασαν προηγουμένως οι συγγετρίες, Αποβλέπουμε ότι θα χρειαστούμε 20 χρόνια μας είπαν για να φτάσουμε σε αποτελέσματα τα οποία ήδη προβλέπονται στον ορίζοντα 2020, 2020. Και μάλιστα σε, σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούμε 40 κιόλα χρόνια για να εφαρμόσουμε και τα προγράμματα της Τρόικα ώστε να μπορέσουμε να πετέχουμε ένα από τους στόχους του ορίζοντα 2020. 40 χρόνια λοιπόν για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Όταν λοιπόν τα ακούμε όλα αυτά, πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Εντάξει, υπάρχουν αιτία πολιτικά, μακροοικονομικά. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Από την Οικονομική Νομισματική Ένωση πήγαμε σε άλλες καταστάσεις. Είχαμε επίσης και τα ευρωπαϊκά εξάμεινα. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας άμεσος συσχετισμός μεταξύ πολιτικών και ιδεολογικών πολιτικών της Ένωσης αφενός και αφετέρου της πραγματικότητας, της πραγματικότητας της καθημερινής που αποτελεί ακριβώς ε, επίπτωση αυτών των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πεμέντα. Τέλος, ο κ. Ορτασούν εκ μέρους των βουλευτών. Πρώτα ευχαριστώ πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω τις ε, τρεις εισηγήτριες που μας ε, παρουσίασαν στοιχεία τα οποία νομίζω είναι πραγματικά καινοτόμα και θα πρέπει να τα αναλύσουμε περαιτέρω ιδιαίτερα αυτά που ακούσαμε στην πρώτη εισήγηση για τον αριθμό των γυναικών που δεν μπαίνουν στην αγορά εργασίας για, οικογενειακούς λόγους Βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει αυξηθεί σε κάποιες χώρες και μας ανησυχεί και στην ομάδα μου. Βλέπουμε ότι αυτή η τάση έχει να κάνει με μια πολιτική που οφείλεται σε μια αποχώρηση από τις δημόσιες υπηρεσίες στην δημόσια ζωή και αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες όσον αφορά την παρουσία τους στην αγορά εργασία και την δυνατότητα που έχουν να έχουν κάποια εισοδήματα από την εργασία τους. Αυτό λοιπόν αντανακλά νομίζω μια πολύ σημαντική κατάσταση και στην έκθεσή μα θα πρέπει ακριβώ να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Και συμμερίζουμε απόλυτα και αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο, δηλαδή για το ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένου στόχου ε, ισότητα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν συζητήσαμε εδώ το εξάμεινο στην Επιτροπή ισότητα, επιμείναμε ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και νομίζω επίση ότι θα έχουμε και εκθέσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά θέματα όπως ας πούμε μερική απασχόληση που όλο και περισσότερο φαίνεται να αφορά την ε, απασχόληση των γυναικών και άλλες προβληματικές γιατί όταν έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε χώρες ε, μέλη Αυτέ οι μεταρρυθμίσεις κυρίω αφορούσαν και επιβάρνα τη μερική απασχόληση που ήταν κυρίω απασχόληση των γυναικών και αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Έχουμε στοιχεία επίση και δημογραφικά. Η τάση δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στι χώρε όπου είχαμε προγράμματα προσαρμογής, εκεί έχουμε την απασχόληση των γυναικών κατά 70%. Αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει ω στοιχείο. Και σχετίζεται με αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή όταν εμεί κάνουμε συστάσει πολιτική στι χώρε μέλη, αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν γίνεται να τα θεωρούμε δεδομένα και εύλογα όλα αυτά, γιατί είναι στοιχεία που αποκαλύπτουν μια ανησυχητική κατάσταση. Στι παρουσιάσει λοιπόν νομίζω ότι μα δώσατε σημαντικέ πληροφορίε, σημαντικό περιεχόμενο, παρόλο που η κυρία Κλικέ, αυτά που είπε δεν σχετίζονται άμεσα με την εισήγησή μα, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω παρόλα αυτά γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Ορτάζουν για τώρα ε, να ολοκληρώσουμε την ακρόση. Έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά το πρόγραμμα μα. Πάντω μπορεί να λέτε το λόγο. Τρία λεπτά ο καθένα. Και οι προσκεκλημένοι μας βέβαια θα λάβουν το λόγο για να απαντήσουν στα όσα ε, έχουν ερωτηθεί η κυρία Λάγκο, πρώτη. Το θέμα της απασχόλησης, τι γίνεται με τη μερική απασχόληση και όχι μόνο για να δούμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κάποια σύμβαση εργασίας που να εξασφαλίζει αποδοτικότητα στην κοινωνία και να εξασφαλίζει και αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν τα αναφέρω αυτό, αλλά τα έχουμε συζητήσει. Αναλύσαμε τις αιτίε. Πρόκειται για δίκτυ. Μιλούμε για ανατομία που κυριαρχούν οι γυναίκες και η αμοιβή εργασία είναι χαμηλότερη και κάπου αλλού που είναι το αντίθετο. Οπότε αυτό λάβετε υπόψη. Ε, τελικά ο δείκτης που μετέρχεται κανείς είναι η απασχόληση. Άρα το πώς γίνεται ο υπολογισμός είναι κάτι που εμπεριέχει πολλές μεταβλητές. Οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα, τα εισοδήματα και προκύπτει το μισθολογικό ε, χάσμα. Δεν λέμε ότι είναι τελείω λάθο αυτό ο υπολογισμό. Είναι κάποιο από του υπολογισμού γιατί ακριβώ η αγορά εργασία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε δηλαδή να μετρήσουμε από εκεί το αν αξιοποιούνται οι δυνατότητέ μα. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναλύσουμε περισσότερο ει βάθο τι γίνεται στον στην παιδεία, τι γίνεται ε, σχέση το ένα φύλλο σχέση με το άλλο, γιατί οι γυναίκες πάνε σε συγκεκριμένου τομεί όπου εκεί δεν κερδίζουν ακριβά και όταν ε, δεν κερδίζουν αρκετά και όταν το συνειδητοποιήσουν είναι τότε αργά και δεν πάνε αλλού που κυριαρχούν οι άντρες. Η απασχόληση είναι ένα κριτήριο, σύμφωνοι. Αλλά ίσως θα πρέπει και πάλι να δούμε στόχους που προσυδειάζουν στο κάθε φύλλο. Τέλος πάντων, να δούμε τις αιτίες, να δούμε τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, πώς μπορεί να υπάρξει νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος επ' αυτού. Ναι, ναι, ναι, δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό το δίκτυο, αυτό το κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Λέγκεμπερ και τώρα έχει το λόγο υπομένη προσκεκλημένη μας. Ε, ευχαριστούμε πρώτα πρώτα όλους όσοι έλαβαν τον λόγο ε, χαίρομαι που καταλάβατε που πήρατε το μήνυμα νομίζω ότι ε, φάνηκε το πόσο αυτά τα κριτήρια που αναφέραμε είναι χρήσιμα σε πόσα μέτωπα λέει η κυρία Μπέτιο δεν είχα το χρόνο να σας τα πω δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο όμως. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι οι αιτίε είναι μόνο μακροοικονομικές. Αλλά λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Αυτό που έχω να σας τονίσω είναι το εξής. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι σίγουρη αν θα έπρεπε να το αναφέρω στην ε, εισήγησή μου ή να το πούμε τώρα. Πολλές φορές για τις νεαρές γυναίκες τα πράγματα διαφέρουν σε σχέση με τις μεγαλύτερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα εκεί και έχουμε πολλά είδη συμβάσεων εργασίας. Διαφορετική οργάνωση της εργασίας, ο ελεύθερος χρόνος, ε, η αμοιβόμενη εργασία, πολλά πολλά ποικίλουν. Δεν υπάρχει κάτι το στάνταρ. Και το σημαντικό εδώ είναι το κατά πόσον η ισότητα των φύλων είναι κάτι το οποίο το ασπάζονται όχι μόνο οι γυναίκες μιας παλιότερης γενιάς, αλλά και οι νεαρές και οι νέες γυναίκες. Δηλαδή, ε, μέσα σε αυτή την ερευστή ώρα εργασίας λαμβάνει υπόψη το τι τους δίνει μια αξιοπρεπή διαβίωση ρευστή αγορά εργασία, πάει να πει ότι πάρα πολλά συμβαίνουν. Μεγάλη κινητικότητα, μεγάλε διαφορέ, μεγάλη ποικιλία. Και βέβαια πολλά προβλήματα και πολλέ δυσκολίε. Δεν ξέρω εάν σα τα είπα ώστε να τα καταλάβετε, αλλά νομίζω ότι εδώ το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει και αυτό να εξετάσει. Τι γίνεται με τις νεαρές γυναίκες αγορά και τις προκλήσεις, τα προβλήματά τους. Δεν νομίζω ότι ε, απασχολούμαστε αρκετά με αυτό. Κύριε Μπέτιο, σας ευχαριστώ. Και ε, τελευταία, αλλά με τον λόγο, κυρία Κλίνγκε. Δεν ρωτήσα τίποτα για τη δική μου σύγχυση, αλλά ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα είναι σύμμαχός μας. Ακριβώς για την ε, ένταξη των θεμάτων των γυναικών στην επεξεργασία της αξιολόγησης όπως κάνουμε. Και για την επόμενη φάση του προγράμματος ε, Horizon 18 με 20. Η πρόταση ευχαριστούμε πολύ για τις εισηγήσεις σας, για τα όσα μας εξηγήσατε. Νομίζω ότι η εισήγηση και η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Έτσι τώρα έχουμε Οι ιδέες που θα μας βοηθήσουν στο έργο μας, δηλαδή να συντάξουμε την έκθεσή μας. Σας ευχαριστούμε και τις τρεις που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που συζητήσατε μαζί μας τα θέματα. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Δίλεπτο διάλειμμα. Dear colleagues, we will start. Please take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε, παρακαλώ, καθίστε. Συνεχίζουμε με την ημέρα διάταξη και περνούμε στο έκτο σημείο της ημέρας διάταξης που είναι η συζήτηση όσον αφορά την ε, έκθεση για την ισότητα των φύλων όσον αφορά την ψυχική και πνευματική υγεία. Κυρία Μπεθέρα είναι η συγγήτρια. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες αρχικές συζητήσεις. Οπότε θα λάβει το λόγο τώρα η συγγήτρια για να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ συνόδελφε και πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι από τότε που κάναμε την πρώτη συνάντηση εκεί όπου συζητήσαμε για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τους κοιόδες από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και υπήρχε πνεύμα συνενετικό, επικοδομητικό οπότε καταρχήν τα πράγματα είναι βέβαια δύσκολα, είναι περίπλοκα και προσπαθούμε τώρα να οριοθετήσουμε τα πράγματα γιατί ακριβώς όπως βλέπετε από τον τίτλο έχουμε θέματα ευρύτατα δεν μπορούμε να είμαστε εξαντλητικοί. Οπότε σίγουρα σε αυτές τις ε, επαφές μας με τους ισοσκιώδες ηγητές συμφωνήσαμε, είπαμε ότι θέλουμε να εμβαθύνουμε στα θέματα της ψυχικής υγείας και επίσης είπαμε ότι η αφετηρία για αυτή την έκθεση δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πρώτα-πρώτα να δώσουμε έναν ορισμό της υγείας. Ο Κόσμος Οργανισμός Υγείας δίνει έναν ε, ορισμό και μιλά για σωματική, ψυχική υγεία και όχι μόνο. Και είπαμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτές οι διάφορες πτυχές για το πώς αντιλαμβανόμαστε την υγεία. Να δούμε επίσης το την αρμοδιότητα της Ένωσης να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οπότε εκεί θα εστιαστούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έτσι να δούμε πού απαιτείται να αναλυφθεί δράση, να δούμε τι δυσμενείς διακρίσεις υπάρχουν, που υπάρχει ανισότητα στο ε, πρόσβαση που είναι και στην υγεία όταν έχουν ιδιαίτερες ε, ανάγκες, ιδίως για την ψυχική υγεία. Ε, επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, τι θα πρέπει να θεωρηθεί ψυχική υγεία των γυναικών. Έχουμε βέβαια και το θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών, τα θέματα της ε, αναπαραγωγικής ε, υγείας, γιατί εδώ έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία προσυδειάζουν περισσότερο στις γυναίκες. Είναι θέματα που πλήσουν, που αφορούν μόνο τις γυναίκες ή κυρίως αυτές. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα καλύπτουν οι υπηρεσίες υγείας αυτές τις παθήσεις ας πούμε. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ε, ψυχική κυρίως υγεία την προστασία θα υπάρχει από τις υπηρεσίες υγείας γιατί υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ομάδες γυναικών που έχουν συγκεκριμένα ε, θέματα και, και ανάγκες όπως οι γυναίκες που ζητούν άσυλο. Έχουμε επίσης και κάποιες πρωτοβουλίες για αυτά τα θέματα που βοηθούν. Κάποιες τροπολογίες λένε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάθλιψη που αφορά ε, πολλές φάσεις και πριν και μετά τον τοκετό επίσης άλλες περιπτώσεις, άλλε αρρώστιες ε, κάποια προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος ενδομητρίωση, αυτοκτονία. Μιλάμε για φαινόμενα τώρα, όχι για αρρώστιες. Είναι μια κατάληξη κάποια συμπεριφορά που δεν καλύπτεται αρκετά από τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την ε, δημόσια ψυχική υγεία. Επίσης έχουμε και τον άλλο άξονα της έκθεσης, την κλινική έρευνα γιατί θα πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ότι οι κλινικές δοκιμές γίνονται χωρίς δυσμενείς διακρίσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνεται 50-50, δίκαια. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία, στατιστικά δεδομένα συμμετοχή των γυναικών, επομένως ισότιμα σε αυτές τις κλινικές δοκιμές. Χρειάζεται να δούμε τι γίνεται με την έγκριση, με την ιδιωτοθεσία για τα φάρμακα. Θα πρέπει να υπάρχουν εξηγήσει όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, γιατί υπάρχουν πάντοτε ε, επιπτώσεις από αυτές τις δοκιμές, παρενέργειες. Άρα, ισότητα στις δοκιμές και θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να δώσει κατευθυντήριες γραμμές που να πιάνουν τόπο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας κυρία Μπεθέρα. Τώρα θα περάσουμε στις ομάδες. Η κυρία Κολόνσκα που αντικαθιστά την κυρία Σταράς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Θα αντικαθεστήσω τη συνάδελφό μου κυρία Έστρα, η οποία λυπάται που δεν μπορούσε να είναι εδώ για την συνάντηση της Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο μου ζήτησα να διαβάσω μερικά σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Πιστεύει ότι δυστυχώς ε, το ε, ποσοστό αυτό απουσιάζει το περιεχόμενο ε, ξεπερνά τις δικαιοδοσίες της ΦΕΜ και ε, υπάγεται στις δικαιοδοσίες της ΕΝΒΗ όπως είναι στις παραγράφους 18, 20 και 21. Επί επίσης υπάρχουν ε, μερικά ε, ζητήματα όσον αφορά τις αμβλώσεις ε, και την προογική υγεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετα όπως αναφέραμε στις κάποιες τέσσερις παράγραφοι δεν ε, δεν αρμόσουν στη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ευρωπαϊκή ε, Συμφωνία για την ψυχική υγεία του 2008, την κοινή δράση για την ψυχική υγεία και ευημερία των Ευρωπαίων 2013-2016, ούτε και την ε, πράσινη βίβλο που εξεδόθη το 2015. Επίσης, η έκθεση δεν αναφέρεται σε ζητήματα όπως είναι, για παράδειγμα, η εκπαίδευση ε, των επαγγελματιών υγείας, ε, καθώς επίσης ε, και την εκπαίδευση για την για τις κλινικές δοκιμές καθώς επίσης και τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου ε, για την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω προτείνει κάποιες τροπολογίες ε, και είναι ανοιχτή να δεχτεί ε, προτάσεις από άλλες πολιτικές μου ομάδες για να βελτιώσουμε την τελική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κολόντσκα. Περνάμε στην κυρία Ward. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το προσχέδιο το οποίο έχουμε δει εμεί είναι ακόμα πολύ γενικό. Αναφέρεται σε κάποια ζητήματα για την υγεία των γυναικών. Όμως θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Πέατρη και το γραφείο της και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά για να ε, ε, εργαστούμε πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο αφορά ένα πολύπλοκο ζήτημα. Θα ήθελαμε όμως να εισάγουμε κάποια σημαντικά ζητήματα για την ψυχική υγεία. Θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση ότι οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν την στρατηγική ε, για την ψυχική υγεία και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία και γίνονται διάφορες δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ε, και πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν τη συγκεκριμένη έκθεση λόγω αυτού του γεγονότος γι' αυτό το λόγο μας ε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω μας. Θα ήθελα να πω ότι πρώτον ε, μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση ε, που συμπεριλαμβάνει ψυχοκοινωνικούς παράγοντες ε, που επηρεάζουν την υγεία μας. Όλα αυτά βοηθούν στην αντιμετώπιση των, ε, φιλοτικών, των ανισοτήτων φύλων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια, την κατάθλιψη ε, στα έφηβα κορίτσια αλλά και σε μεγαλύτερες γυναίκες. Όλο αυτό απαιτεί να έχουμε μια γενικότερη προσέγγιση για να μπορέσουμε να ε, αναφερθούμε στα ζητήματα ψυχικής υγείας ανθρώπων κάθε ηλικίας και θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσέγγιση στα παιδιά και τους νέους θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ε, καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και το στίγμα σχετικά με την ψυχική υγεία. Και υπάρχουν ήδη καλές πρακτικές ε, σε διάφορους οργανισμούς ε, της κοινωνίας των πολιτών. Τα αγόρια και οι άνδρες επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ε, και εν μέρει εξαιτίας των ε, στερεοτύπων ε, και αυτό οφείλεται στην κατάχρηση ουσιών και στα υψηλά ποσοστά ε, αυτοκτονιών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το ξεχνάμε αυτό στην Επιτροπή μας. Επίσης υπάρχουν και άλλες ζητήματα όπως η ανησυχία για την ψυχική υγεία των μεταναστών και των προσφύγων γυναικών ε, όπως επίσης και γυναίκες με αναπηρία και γυναίκες που παρέχουν φροντίδα. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, το γεγονός ότι τα φάρμακα δεν δοκιμάζονται τόσο συχνά σε γυναίκες, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ζωή τους. Η έρευνα από την Χάνη να περιλαμβάνει το φύλλο ως έναν παράγοντα στην όλη διαδικασία και οι γυναίκες είναι υπο, υποεκπροσωπούνται στις δοκιμές και νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εκτιμώ λοιπόν το έργο που κάνει η Μπέατρης πάνω σε αυτό ή ο αναθεωρισμένος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014 ορίζει ότι θα πρέπει το φύλλο να συμπεριλαμβάνεται στις δοκιμές, όμως γνωρίζουμε ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις καρδιακές ασθένειες, καθώς επίσης και στη θεραπεία για εγκεφαλικά. Καλό λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας μαζί με τους Κιώδης για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γουρτ, και τώρα πάμε στην κυρία Πιόρκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια για το έργο της. Νομίζω ότι πολλά από τα όσα έχουμε συζητήσει συμπεριλαμβάνονται ισότητα, τα δικαιώματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, ε, ε, το ζήτημα των ε, προσφύγων ε, γυναικών, η ενδομητρίωση και ιδιαίτερο το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για να θέσει την υγεία ψυχική και σωματική των γυναικών στην σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, για να ενισχύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συζητήσουμε για τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και ε, τα, ε, τις ασθένειες από τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ζητήματα κούρασης, ε, την υγεία των νέων κοριτσιών, ε, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την σεξουαλική βία, τους, τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔ. Ε, ανθρώπους με αναπηρία και επίσης ε, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο των, ε, των υπαλλήλων του τομία υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπιόρκ. Ολοκλήρωσαμε το, τον γύρο των ερωτήσεων και παραμβάσεων. Κυρία Μπεθέρα, θέλετε μήπως κάτι να σχολιάσετε μετά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Είναι σύντομα να ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή τους και τον ενθουσιασμό τους για αυτό το θέμα. Όπως είπε και η Γιούλη, η καλύτερη ημέρα είναι σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συνεργασίας και κατανόησης θα ήθελα να έχουμε κάτι κατά νου ότι στο τομέα της ψυχικής υγείας δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τίποτα. Όλα μετράνε για την ψυχική υγεία και την ψυχική ευημερία των γυναικών. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί και περιεκτικοί όταν προσεγγίζουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα που το γνωρίζουμε άμεσα σε προσωπικό επίπεδο όλοι μας όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Όταν πάμε σε ένα γιατρό, όταν θα πρέπει να πάρουμε ένα φάρμακο. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν, ας πούμε, κάνουμε χείριση και για τα δικαιώματα αναπαραγωγής. θα ήθελα να μιλήσουμε και για το δικαίωμα στην άμβλωση. Όπως είπε και η συνάδελφος που αντικαθιστά από το ΕΛΚ την κυρία Σαράς. Νομίζω ότι εδώ καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε νόμιμες δομές και υπηρεσίες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με την συναισθηματική, φυσική και ψυχολογική σταθερότητα των γυναικών. Ιδιαίτερα έχουμε να κάνουμε εγκυμοσύνες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ε, φυσική για των γυναικών και κυρίως οι αμβλώσεις βέβαια, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε όλοι οι εμπειρογνώμονες, όλοι οι ειδικοί του κόσμου και είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί πια. Οπότε, μια και μιλάμε στην έκθεση για ψυχική υγεία και τις διακρίσεις των γυναικών, εις βάση των γυναικών στην πρόσβαση, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Δηλαδή να μην υπάρχει πρόσβαση σε ένα κομμάτι των υποδομών υγεία, στα οποία οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση. Ίσως να διαφωνήσουμε στην διατύπωση στις λέξεις, αλλά νομίζω συμφωνούμε επί της ουσίας. Μιλάμε για δικαίωμα αναπαραγωγής. Μιλάμε για τα δικαιώματα που αφορούν την φυσική και την πνευματική ψυχική υγεία των γυναικών. Οπότε θα ήταν καλό να βρούμε έτσι ένα σημείο επαφής, επικοδομητικό και χρήσιμο για τις γυναίκες της Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω αυτό που είδαμε στην Πολωνία πρόσφατα. Δεν είναι κάτι δηλαδή το θεωρητικό. Είναι κάτι το οποίο είναι απτό, υπάρχει, έχει εμφανιστεί ήδη. Κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν διασφαλισμένο, επειδή περιλαμβάνεται στις διεθνείς συνθήκες, στις συμβάσεις, στις συμφωνίες. Θεωρούσαμε ότι ήταν διασφαλισμένο. Δεν χρειάζεται να το κάθε φορά και όμως δεν είναι έτσι. Κάτι άλλο που είπε η Γιούλη για συγκεκριμένα περιστατικά πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαστούμε. Νομίζω ότι υπάρχει υπο, υποεκπροσώπηση των γυναικών στις, στις κλινικές δοκιμές. Οπότε η έρευνα δεν μπορεί de facto να είναι καλή και δεν μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Γιατί ο πληθυσμό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η έρευνα, η οποία σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτείται από πόρου τη Ένωση θα πρέπει βεβαίω να παρουσιάζει την πραγματικότητα. Και σε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση που είπε η συνάδελφος Μπιόρκ. Είναι αλήθεια ότι στο χώρο εργασίας υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις που έχουν να κάνουν ακριβώς με την ε, ψυχική υγεία των ε, γενικών. Δεν μιλάμε μόνο για την όχληση, τη σεξουαλική ή άλλα φαινόμενα ή την εργασιακή ας ανασφάλεια επειδή οι γυναίκες ας πούμε δεν μπορούν να φτάσουν σε αξιοπρεπή όρια διαβίωσης με το εισόδημά τους, με το μισθό τους σε σχέση με τους άντρες αδέλφους τους. Όταν μιλάμε για ψυχική υγεία το ξαναλέω και επιμένω. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ τον ορισμό που δίνουν οι ειδικοί και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτά που λέει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Δηλαδή να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Γιατί η ψυχική υγεία αφορά όλε τι πτυχέ τη ζωή μα. Και οι κλινικές έρευνες είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν σωστά και πρέπει να ζητήσουμε και ευθύνε όσον αφορά κάποια φάρμακα, αλλά να συζητήσουμε ακριβώς και το θέμα της χρηματοδότησης των ερευνών εκ μέρους της Ένωσης για κονδύλια για τα οποία δεν υπάρχει αντίκρισμα όσον αφορά τις τιμές στα φάρμακα. Θα κάνουμε λοιπόν μια έκθεση η οποία θα βασίζεται στις συνθήκες και στις συμφωνίες γιατί είναι τόσο σημαντικές και τόσο πολλές οι που αν συζητήσουμε και συμφωνήσουμε τουλάχιστον για του βασικού πυλώνε, θα κάνουμε κάτι ουσιώδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπεθέρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι 17 Οκτώβρη στις 17.05 το απόγευμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξη τώρα που αφορά την κατάσταση των γυναικών προσφύγων στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας θα κάνει μια αποστολή στην Ελλάδα για να γνωρίσει από κοντά την κατάσταση που αφορά αυτές τις γυναίκες πρόσφυγες. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και καιρό. Είχαμε την έκθεση Honeyball. Είχαμε και την Παγκοσμία ημέρα της γυναίκας στην οποία επικεντρωθήκαμε στις γυναίκες πρόσφυγες. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε επιτόπου την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτέ οι γυναίκε στην επικράτεια τη Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την επίσκεψη στην Ελλάδα. Και προηγουμένω θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό για μας να έχουμε έτσι μια εικόνα πιο άμεση, πιο κοντινή. Γι' αυτό ακριβώς θεωρήσαμε καλό να καλέσουμε την ε, κυρία Κούβελα, η Γενική Γραμματέα Ισότητας, που γνωρίζει βεβαίως όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενική κατάσταση των γενικών προσφύγων και τα θέματα που αφορούν επίσης την ε, βοήθεια στα θύματα, την καταπολέμηση της ε, λαθρεμπορίου, μάλλον της διακίνησης γυναικών. Όλα αυτά σε σχέση με την επίσκεψή μας στις 3 και 4 Νοέμβρη. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Κούβελα που είχε την ευγένεια να έρθει εδώ σήμερα το απόγευμα και θα της δώσω το λόγο για να κάνει την πρώτη σε εισαγωγική παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Ε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με τη σημερινή μου παρουσία εδώ στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση της προσβητικής κρίσης, η οποία πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά. Όπως γνωρίζετε, εν μέσω μεγάλων οικονομικών δυσκολιών, ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει και τη μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης της προσβυγικής και της μεταναστευτικής κρίσης. Μια πρόκληση παγκόσμια, την οποία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο συλλογικά και με βάση τις αξίες μας, χωρίς να χάνουμε την ανθρωπιά μας, η οποία δεν τίθεται υπό όρους. Από τη στιγμή που τα βόρεια σύνορά μας έκλεισαν, λόγω μονομερών ενεργειών άλλων χωρών, περίπου 60.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σήμερα στην Ελλάδα. Η άμεση αυτή ξενοφοβική αντίδραση λειτουργήσε πολύ συχνά όχι και έλεσμα να θυσιαστεί το διεθνές δίκαιο και να επαναπροωθούνται πρόσφυγες, ακόμα και διακινδυνεύοντας τις ζωές τους στη θάλασσα. Πολύ συχνά ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου θεωρήθηκε πολυτέλεια και όχι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης. Πολλές φορές ο επιμερισμός της ευθύνης για τους ανθρώπους που επιχειρούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις απορρίφθηκε ως ευθύνη που βαραίνει μόνο τα κράτη πρώτης γραμμής. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συνεκτική, συλλογική απάντηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης με υποστήριξη φυσικά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στην Ευρώπη εργαζόμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μια συμφωνία δύσκολη που έχει οδηγήσει ωστόσο σε δραστική μείωση των ροών και το σημαντικότερο των θανάτων στο Αιγαίο Πέλαγος που έχει αντικαταστήσει την επικίνδυνη διαδρομή του Αιγαίου με μια νόμιμη οδό προς την Ευρώπη. Αλλά χρειάζεται να αναπτύξουμε μια ευρύτερη παγκόσμια στρατηγική ώστε να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση και η ενίσχυση με προσωπικό προς τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής ανθρώπων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, καθώς και η επανακατάσταση και μετακατάσταση των προσφύγων. Να αυξηθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης να αυξηθεί η αστυνόμευση των συνόρων και η συνεργασία των ακτοφυλακών για την εξάλληψη των δικτύων εμπορίας ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, και με σεβασμό στις αξίες και στα θεμελιώδη. Στο πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στις αξίες και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στέκεται αλληλέγγυα και συντονίζει τη δράση της, τις δράσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020 περιλαμβάνονται δράσεις και στόχοι πολιτικής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών που υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις με έμφαση τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγου φύλου πολλαπλασιάζονται και οξύνονται, μέσα και από άλλες μορφές διακρίσεων, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκαταλήψεις, τη μυσαλλοδοξία, την έμφυλη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, χαράσουμε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο παρέμβασης. Συγκροτήσαμε τη Συντονιστική Επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και άλλων συναρμόδιων κομφορέων καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες, θύματα ή ενδυνάμει θύματα βίας και στα παιδιά τους ή σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Έργο της Επιτροπής είναι και η χάραξη του πλαισίου των επιμέρους συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς ή ελληνικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο θέμα του προσφυγικού για την ανάληψη από κοινού δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να αξιοποιηθεί θετικά το δίκτυο των 61 δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που λειτουργούν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα η Συντονιστική Επιτροπή έχει επεξεργαστεί και παραδώσει το σχέδιο ενός πρωτοκόλου συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται η διαδικασία και οι ενέργειες που οφείλουν να κάνουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο στάδιο του εντοπισμού των γυναικών προσφύγων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, στις ανοιχτές δομές προσωρινής υποδοχής και τις ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας, και στην παραπομπή του στα συμβουλευτικά κέντρα ή στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τους ξενώνες φιλοξενίας. Περαιτέρω υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν εφόσον διασφαλιστεί και η διερμηνία ή η διαπολιτισμική μεσολάβηση είναι η εξής. Ασφαλής διανομή στους ξενώνες φιλοξενίας. Σήτηση κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, νομική συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική, δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης που αποσχολούνται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, σε όλες τις δομές δηλαδή που έχουμε, θα μπορούν να συντονίζονται μεταξύ τους για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας ή γυναικών προσφύγων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και συνδρομής. Ενώ παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία των ετοιμάτων φιλοξενίας από ειδική βάση δεδομένων που ήδη υπάρχει για τις περιπτώσεις γυναικών θυμάτων βίας και τώρα θα αποκτήσει ειδική καταγραφή για τις ωφελούμενες γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Περαιτέρω θα προχωρήσουμε στην ενημέρωση όλου του προσωπικού για το πλαίσιο διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και στήριξης των ωφελουμένων γυναικών, προσφύγων και των παιδιών τους, στο σχεδιασμό επιμόρφωσης κατάρτισης για τις διαδικασίες ασύλου, μετεκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης, σε βασικές κατευθύριες οδηγίες για τη διαδικασία προστασίας γυναικών προσφύγων, θυμάτων ή ενδυνάμει θυμάτων βίας, σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ήδη σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες εργαζόμαστε από κοινού στην επικαιροποίηση των κατευθύνων οδηγιών για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα έχουν ήδη μεταφραστεί στις γλώσσες που ομιλούν οι γυναίκες πρόσφυγες τα έντυπα και ο κανονισμός λειτουργίας των ξενών φιλοξενίας και ετοιμάζεται και ειδικό φυλάδιο που θα απευθύνεται στις ίδιες για να ενημερωθούν και τις υπηρεσίες που μπορούν να τις παρασχεθούν. Επίσης, σε συνεργασία με την UN Women θα διοργανώσουμε δύο συνέδρια, όπου όλο το προσωπικό που δρά στο πεδίο θα επιμορφωθεί στις πολιτισμικές διαφορές και τη διαδικασία ασύλου και παροχής διεθνούς προστασίας, ενώ θα γίνει και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας περιέγραψα συνοπτικά τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό μας, ενώ αρκετά σύντομα θα συντονίσουμε τη δράση μας και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, στην κατεύθυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων, που θα συνδύνουν στην κοινωνική ένταξη των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας ξεκινάει τη λειτουργία δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων με στόχο να καλυφθούν φέτος περίπου 22.000 παιδιά. Ήδη έχουν αρχίσει να πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία προσφυγόπουλα. Ενώ μέσα από το νέο νόμο που έχει προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία θα αναζητήσουμε δυνατότητες ώστε οι γυναίκες να μπορούν να αποσχοληθούν ή και να δημιουργήσουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού ή τις Περιφέρειες μπορούν να διοργανωθούν πολιτιστικές εξορμήσεις των γυναικών προσφύγων και επαφή τους με το πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας που τις έχει αγκαλιάσει και τις έχει υποδεχτεί. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θεωρούμε κρίσιμη τη συμβολή της δικής σας Επιτροπής για την ανάδειξη του παγκόσμιου χαρακτήρα της προσφυγικής κρίσης και την αποκοινού ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που θα στηρίζονται στις κοινέ αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας, ώστε να περιθωριοποιηθεί και αποφευχθεί ο κίνδυνος της μυσαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούβελα για την εισήγησή σας. Και τώρα θα έχουμε έναν ε, γύρο ερωταπαντήσεων. Πρώτη κυρία Μπιόρκ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε την κυρία Κούβελα που ήρθε στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αποφασίσαμε να ασχολούμε με αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και να δούμε τι βελτιώσεις μπορεί να γίνουν υπέρ των ε, προσφύγων, των μεταναστών. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και με έχει εντυπωσιάσει το έργο σας, κυρία Κούβελα, και λαμβάνοντας υπόψη το, τη συγκυρία στην Ελλάδα. Εγώ προέρχομαι από την Σουηδία. Και εμείς έχουμε δεχθεί περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες από άλλες χώρες. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και περισσότερους, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως ε, δεν μας έχει πληθεί μας κάποιο παράλογο πρόγραμμα. Ε, έχουμε συστήματα υγείας και συστήματα εκπαιδευτικά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες πρόσφυγες. Θέλουμε να περιορίσουμε ρατσισμό και ξενοφοβία. Βέβαια, Το πρόβλημα αυτό υπάρχει παντού, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ε, όλοι όσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να προωθήσουν το θεματολόγιο του οι ρατσιστέ. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε αυτέ τι δυνάμει. Οπότε και για τη δουλειά σε αυτό το μέτωπο σα ε, ευχαριστούμε. Έχω δύο παρατηρήσει και δύο ερωτήσει να σα κάνω. Μα αναφέρετε τι 60.000 πρόσφυγες. Αυτοί που τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν μπορούν να φύγουν, μια που τόσες χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα τους. Πόσοι από αυτές τις 60.000 είναι γυναίκες και ανήλικοι, μας είπατε για 32.000, αν δεν κάνω λάθος. 32.000 ανήλικοι που πρόκειται να πλαισιωθούν από τα ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι υπέροχο. Αν λάβει κανείς υπόψη τη δύσκολη συγκυρία της παιδεία Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο στην Σουηδία. Οπότε από τι 60.000 πόσοι είναι ανήλικοι και πόσε γυναίκε παρακαλώ. Επίση, πέστε μα, τι θα συνιστούσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα περιμένατε από εμά. Δύο φορές έχω ταξιδέψει στην ε, Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα, όταν είχαμε τον διάδρομο, τον ανθρωπιστικό, τότε που άνοιξε αυτός ο διάδρομος μέσω Σερβίας προς Γερμανία, και είχαμε τότε σχετικές συνθήκες ασφάλειας, σχετικής ασφάλειας τέλος πάντων. Αργότερα κλείσαν τα σύνορα και τότε πήγα, πήγα στην ε, ε, Λέσβο και συνάντησα πολλές γυναίκες, ήταν πολλές εκεί γυναίκες και τα παιδιά που ήταν αποκλεισμένα ε, ούτως πίν στο νησί και περίμεναν να πάνε προς Γερμανία, Σουηδία, όπου τους περίμεναν οι οικογένειές τους. Όπως λέει ο κανονισμός του Δουβλίνου, δικαιούνται να μεταβούν σε Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πρόκειται για παρένωση οικογενειών. Γιατί δεν υλοποιούνται αυτά που προβλέπει ο κανονισμός. Βρίσκονται τώρα έξι μήνες, ένα χρόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να πάνε στις οικογένειε τους. Τι να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Επίση, για πετε μου και τη χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση προς την Ελλάδα, αλλά δεν περνάει από την κυβέρνηση. Η χρηματοδότηση αυτή ε, πάει σε ΜΚΟ, πάει ε, στις οργανώσεις, στην οργάνωση τέλο πάντων του, του ΟΗΕ και τελικά βοηθάει όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων. Δεν θα πρέπει κάπως να οργανωθεί καλύτερα το θέμα για να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ και η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κοβέλα για την παρουσίασή της. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε εν ώψη της αποστολής μας στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα της συμφωνίας με την Τουρκία γιατί δεν είναι το κατάλληλο μέρος εδώ. Όμως θα ήθελα να πω ως Πορτογαλίδα ότι κατανοώ πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την λιτότητα. Δεν χρειάστηκε μόνο δηλαδή να υποστεί τη λιτότητα, αλλά μετά βρέθηκε μπροστά σε αυτή την τεράστια μεταναστευτική ροή και χρειάστηκε να διαχειριστεί όλο αυτόν τον κόσμο. Και απέδειξε ακριβώς το τι εννοούμε με ανθρωπισμό εμείς οι Ευρωπαίοι. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ώστε να προσπαθήσουμε έτσι να ερευνήσουμε το βαθμό εκπαίδευση αυτών των ατόμων που εισέρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνετε κάποιο είδος αποτίμηση ή αξιολόγηση των διπλωμάτων που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μίλησαμε και για κατάρτιση για τις γυναίκες πρόσφυγες. Αυτό το κατάρτισης πώς το έχετε διαρθρώσει, πώς το έχετε σχεδιάσει. Και καταλήγοντας να πω το εξής. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι, σημαίνει, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την κατανομή των προσφύγων σε άλλε χώρε όπω και η Πορτογαλία. Εμεί συνεχίζουμε να περιμένουμε του προσφυγέ. Έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των προσφύγων που είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ενώ φτάνουν με το σταγονόμετρο αντίθετα. Ξέρω ότι υπήρξαν άμεσε επαφέ με την Ελλάδα, με την Ιταλία κτλ. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει αυτή η συστηματική καθυστέρηση. Τη στιγμή που έχουμε μακρά παράδοση ενσωμάτωση στη χώρα μα προσφύγων και ξένων στι κοινωνίε μα. Τελευταία ερώτηση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ αναφέρομαι και στις ε, χρηματικές ενισχύσεις, τα κονδύλια από την Κομισιόν σε επίπεδο όλων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ η κυρία Μπεθέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Κούβελα. Όλοι πραγματικά έχουμε μεγάλη επιθυμία να κάνουμε αυτό το ταξίδι για να δούμε την κατάσταση από κοντά. Οι συντρόφισσες αναφέρθηκαν επανειλημμένως σε κάποια ζητήματα από τα κονδύλια κλπ. Να σας ρωτήσω μόνο επιπλέον το εξής. Εσείς σε αυτόν τον άνθρωπο του Ηρακλή που αντιμετωπίζετε πώς θα βοηθήσει η υλοποίηση της ειδική υπηρεσίας των συνόρων με πόρους ανθρώπινους και υλικούς, ώστε να σας βοηθήσουν να συντονίσετε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την άφηξη και τη μετώπιση όλων αυτών των ατόμων που φτάνουν στην επικράτειά μας και ιδιαίτερα στην δική σας επικράτεια. Και σε σχέση με την τωρινή κατάσταση που αφορά τους χώρους υποδοχής όπου υπάρχουν πάνω από 60.000 άτομα, πάνω από το ίμιση γυναίκε και παιδιά. Πρόσφατα νομίζω, τώρα το Σαββατοκύριακο, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε σχέση με τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των χώρων υποδοχή. Βλέπω ότι κάποιοι χώροι είναι παλιέ τουριστικέ υποδομέ όπου φιλοξενούνται τα άτομα αυτά υπό συνθήκε αρκετά αποδεκτέ, αρκετά καλέ, αλλά Δυστυχώ η ζωή αυτών των ατόμων συνίσταται στο, στην αναμονή. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι χρειάζεται το τάδε ή το δίνα, γιατί εντάξει υπάρχουν παντανάκες, αλλά κυρίω τι απάντηση, πώ θα ανταποκριθούμε εμεί στην ανάγκη για το μέλλον αυτών των ατόμων που ήδη βρίσκονται εκεί στην Ελλάδα, ώστε να διοργανώσουν, να οργανώσουν, να φτιάξουν τη ζωή του τέλο πάντων και να μην έχουν έτσι, αυτή την κατάσταση σε μια παθητική και αδρανή αναμονή που τους φτύρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Κούβελα για να απαντήσει στα ερωτήματα, θα ήθελα να πω και εγώ ως Πρόεδρος ότι την ευχαριστώ για την παρουσία της, αλλά και για την προσπάθεια που ξέρουμε ότι καταβάλλεται για την διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης την οποία έχουμε συνηθίσει επανειλημμένως εδώ στο Κοινοβούλιο και εδώ στην Επιτροπή μας ζητώντας και διεκδικώντας ρόλο για τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης όταν μιλάμε για πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε λοιπόν εργαλεία ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγες στην Ελλάδα, αλλά πρόσφυγες στην Ένωση. Οπότε η απάντηση θα πρέπει να είναι αλληλέγγυα και συνεργατική. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσπάθεια που καταβάλλετε, την τεράστια, και να ξέρετε ότι εδώ στην Επιτροπή μας θα έχετε πάντοτε συμμάχους όταν θα χρειαστεί να διεκδικήσετε περισσότερους πόρους και κονδύλια για τη βοήθεια για τις γυναίκες πρόσφυγες που θεωρούμε ότι είναι οι πιο, τα πιο ευάλωτα άτομα, οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Κύριε Κουβέλα, ευχαριστώ και πάλι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Να σας ε, επισημάνουμε ορισμένα ακόμα στοιχεία. Ε, θέλω να πω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι, πρόσφυγες, γυναίκες και άνδρες και τα παιδιά τους στην Ελλάδα είναι ότι δεν τηρεί τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ποσόστοση. Δηλαδή έχει βγει μια ποσόστοση, όλες οι χώρες της Ευρώπης ανάλογα ε, τη δυνατότητα που έχουν και έχουν δυνατότητα. Δεν είναι υπερβολική, δεν υπερβολική η αριθμή, δεν είναι υπερβολική 60.000 άνθρωποι να φιλοξενηθούν μέσα στην Ευρώπη. Είναι, είναι, είναι μικρό το ποσοστό, είναι μικρό το νούμερο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει θέληση και υπάρχουν και πολιτικές που είναι και ενάντια. Το να κλείνουν τα σύνορα με το έτσι θέλω, με το ε, να γίνονται και δημοψηφίσματα. ευτυχώ αποτύχανε ας πούμε, αυτές οι δυνάμεις. Και δείχνει και μια κατεύθυνση, ας πούμε, που θα πάει η Ευρώπη. Όταν έχει, αν δεν έχουμε ανθρωπισμό στην Ευρώπη, να, ε, να στεκόμαστε αλληλέγγυοι ε, πάνω σε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με πολέμους, με οικονομικές ανισότητες κλπ. Στην ιστορία η ανθρωπότητά μας έχει περάσει πολλές μεταναστευτικές ώρες. Αν δούμε πίσω στην ιστορία, όλες οι χώρες έχουν μετανάστευση. Ας πούμε. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο φυσιολογικό σε, σε παρένθεση, δηλαδή υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του, του αιώνα, ας πούμε. Ε, τώρα βέβαια έτυχε στις δικές μας μέρες, ας πούμε. Και πρέπει εδώ να, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, το πρώτο που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη, να υπάρχει οι μέρη από όλε τι χώρε να πάρουν τον ανάλογο αριθμό προσφύγων που πρέπει, να απεγκλωβιστεί και από την Ελλάδα. Δεύτερο, ένα άλλο θέμα. Ε, ήταν να βοηθηθεί η Ελλάδα με 400 άτομα από όλη την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουν πάει μόνο 19 να βοηθήσουν. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα πρέπει εμείς εσείς εδώ ως ευρωβουλευτές, ευρωβουλεύτες κλπ. να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Πόσοι άντρε, πόσοι γυναίκε, ε, θέλουμε να πούμε ότι έχουμε 22 παιδιά αυτή τη στιγμή που θα βάλουμε σε σχολεία με τι ε, μικρέ μα δυνάμει, αλλά ε, μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Η χρηματοδότηση θα ήταν καλό αντί να πηγαίνει μόνο σε ΜΚΟ, τα περισσότερα χρήματα πάνε σε ΜΚΟ, να δοθούν στο ελληνικό κράτο. Θέλω να σα πω πόσο σημαντική βοήθεια δίνουν απλέ γυναίκε και άντρε στις, ε, στις με πρόσφυγες και στους πρόσφυγες που πάνε σε καθημερινή βάση σε αυτές τις δομές που φιλοξενούνται και προσφέρουν ε, ουσιαστική και καθημερινή βοήθεια πάνω στα καθημερινά προβλήματα που έχουν κυρίως οι γυναίκες. Ε, απλές, απλές βοήθεια, απλή βοήθεια καθημερινή σε πράγματα που λόγω και των δικών τους πολιτιστικών ας πούμε, στοιχείων δεν ξέρουν ε, αυτή η βοήθεια που δίνουν αυτές οι γυναίκες ε, είναι αναντικατάστατη. Ε, όσο αφορά τώρα την ε, εκπαίδευση, δεν μιλήσαμε για κατάρτιση των γυναικών μεταναστριών προσφύγων, ας πούμε, αλλά για να καταρτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό που ασχολείται με αυτό το θέμα, με αυτό το πρόβλημα, ώστε να ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και εδώ θα κάνουμε συνεργασίες και με ΜΚΟ και θα κοιτάξουμε να πάρουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται δηλαδή να εκπαιδευτούν και στα νοσοκομεία οι γιατροί που, και οι νοσοκόμοι που παίρνουν γυναίκες και η αστυνομία να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Ιδίω πρέπει να δούμε πολύ το θέμα της βίας, γιατί αυτές ε, οι γυναίκες ε, έχουν υποστεί ε, βία, ας πούμε. Ε, επίσης αντιμετωπίζουν το θέμα του τράφικινγκ. Αυτά όλα θέλουν μια συνεργασία όλων των φορέων για να μπορέσουμε πρώτα-πρώτα να, την, εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες, να, τις, ε, να εμπιστευτούν και να ανοίξουν την, ε, να το πούν το πρόβλημά τους. Είναι πολύ δύσκολο έτσι. Όταν μια γυναίκα μετανάστρια ε, τρώει ξύλο από το σύζυγό τη και είναι εγκλωβισμένη σε μια ξένη χώρα, δεν έχει που να πάει κλπ. Δύσκολα μπορεί να πει το πρόβλημά τη. α πούμε. Εμείς όμως ε, έχουμε αυτές τις δομέ στη χώρα μας και θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε αυτές οι γυναίκες να μπορούν να, να μιλήσουν. Ε, λοιπόν, ε, επίσης πρέπει να δοθεί, να δοθεί και μια οικονομική δυνατότητα και στη Τουρκία η Τουρκία έχει, μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι η πρώτη χώρα που δέχεται αυτές τις, ε, τους πρόσφυγες. Άρα λοιπόν πρέπει και εκεί να τηρηθεί μια συμφωνία και να δοθεί η χρηματοδότηση. Η δε συμφωνία που κάναμε ε, με, την, ε, με την Τουρκία, ε, πότε έγινε, έγινε όταν κλείσανε τα σύνορα. Κάπω έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα. Αυτά τα μέτρα που πήραμε, αυτή η συμφωνία, ε, ε σας είπα ότι έχει το εξή καλό, ότι σταμάτησαν να πνίγονται πια στι θάλασσε του, του Αιγαίου. Αντίθετα, που έχουμε πρόβλημα τώρα, έχουμε στις ακτές της Ιταλίας, που πνίγεται εκεί ο κόσμος, ας πούμε εντοπίστηκε, ε, ε, μετατέθηκε εκεί το πρόβλημα. Τουλάχιστον από αυτή την άποψη ήταν σωστή αυτή η συμφωνία γιατί σταμάτησε τις, ε, το θάνατο στο Αιγαίο. Δηλαδή έχετε δει όλες αυτές τις σκληρές σκηνές ας πούμε μέσα από την τηλεόραση. Όσοι, έχουν επισκεφτεί και τη χώρα και εδώ οι φίλοι μας από τη Σουηδία ε, έχει μια προσωπική εμπειρία. Ε, εντάξει, μιλάμε για για παράδειγμα, ας πούμε, που δεν τα περίμενε και κανένας να ζήσει. Λοιπόν, ε, χρειάζεται η αλληλεγγύη των γυναικών σε όλη την Ευρώπη σε αυτό. Να, να ενώσουμε τις φωνές μας, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτό το πρόβλημα. Μέσα από την ανθρωπιά μας, μέσα από τη δημοκρατία, μέσα από τις αρχές που έχουν ε, υπερισχύσει τόσα χρόνια στην Ευρώπη και δυστυχώς πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Να μην πάμε πίσω σε αξίες μας. Ε, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποια ερώτηση. Ήθελα να προτείνω επίσης, αν ε, εν ώψη της, ε, θα το έλεγα εδώ στην ε, επικεφαλή της Επιτροπής, μήπως η 8 Μάρτη να είναι μια μέρα αφιερωμένη στην πρόσφυγα γυναίκα. Να σας κάνω μια πρόταση, να σκεφτούμε. Και άλλες δράσεις εν ώψη της 8 Μάρτη. Ε, αυτά. Eh, η πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούβελα. Και όπω είπαμε προηγουμένω, φέτο, το 16 δηλαδή, θα εορταστεί ε, εορτήσει τέλο πάντων στην 8η Μαρτίου η μέρα της γυναίκας και έχουμε την συνάντηση εδώ με γυναίκες πρόσφυγες με βουλευτές από διάφορες χώρες της Ένωσης ενδιαφέρουσα θα είναι η συνάντηση, οπότε και θα προχωρήσει αυτή η δουλειά διακοινοβουλευτικά και με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα. Ελπίζω δε ότι έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε, δηλαδή να ξέρουμε περισσότερο τι γίνεται. Και με την από στην Ελλάδα θα καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται με τις πρόσφυγες. Πάντως σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας τα εξηγήσατε όλα αυτά σήμερα. Και πάλι ευχαριστούμε πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είναι το τελευταίο σημείο για σήμερα. Είναι το θέμα υπαριθμών 8 και αφορά την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Και την έχει αναλάβει η κυρία Μπεθέρα, η οποία και έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ποιο είναι το πνεύμα αυτής της γνωμοδότησης, γιατί θα πρέπει να δούμε πού εστιάζουμε την προσοχή μας. Είναι η βία κατά της γυναίκας. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ε, εκτεταμένο σε όλο τον κόσμο. Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα που αφορά όλες τις χώρες, ε, οριζόντιο μπορούμε να πούμε. Οπότε και αυτό που σας προτείνω είναι να έχουμε αυτό ως άξονα της έκθεσης και επιμέρους στόχοι να είναι το τι κάνει ο ΟΗΕ, τι εργαλεία έχει ο ΟΗΕ για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα, πώς θα υπάρχει πρωτοπορία της ε, γυναίκας για την ειρήνευση, τι γίνεται με την παιδεία και πέρσι άλλωστε είχαμε τη μέρα της γυναίκας και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η εκπαίδευση για τις ε, νεαρές γυναίκες και ανήλικες. Έχουμε εθνικά σχέδια ε, για την υλοποίηση του ψηφίου 13-25 και είπαμε ότι με την ε, εκπαίδευση θα έχουμε χειραφέτηση, θα έχουμε περισσότερη ισότητα και επίσης να λάβετε υπόψη το αν μπορούμε να έχουμε ένα νομοθέτημα διεθνές από πλευράς του ΟΗΕ που να έχει δεσμευτική ισχύ. Να πρόκειται από τον ΟΗΕ λοιπόν και προσπαθούμε εδώ και κάποιο καιρό να ε, δούμε πόσο σημαντικό εργαλείο, πόσο θα το εκμεταλλευτούμε το σύμφωνο της Κωνσταντινούπολης. Να έχουμε πάντως ένα νομοθέτημα εμβέλειας ΟΗΕ, δεσμευτικό για τον έλεγχο των πραγμάτων. Αυτό θα μας βοηθούσε για να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά της γυναίκας σφαιρικά. Αυτά. Ε, ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ κύριε Μπεθέρα, λέει πρόεδρος. Για το Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ε, κάποια ε, πράγματα αντί της κυρίας Γκαμπριέλ για τη συγκεκριμένη έκθεση. Αρχικά θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη που δεν βρίσκεται εδώ, όμως συμμετέχει στην συνάντηση ε, της Επιτροπής ΦΕΜ στην Βαρκελόνη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε ε, την εισηγήτρια ε, για την έκθεση η οποία έχει αρκετά θετικά στοιχεία ε, περιλήφθηκαν ήδη αρκετά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την Επιτροπή ε, ΦΕΜ σε αυτό το προσχέδιο έκθεσης ε, ως εισηγήτρια της EPP. Ε, ε, θα θέλαμε να καταθέσουμε μερικές τροπολογίες για να περιληφθούν κάποια στοιχεία ακόμα. θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα εξ αυτών. Πρώτον, όσον αφορά την χρήση σεξουαλικής βίας ως ε, όπλο πολέμου, επιμένει ε, να συνεχιστεί ε, η καταπολέμηση της έλλειψης δικαιοσύνης και επιθυμούμε την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του δικαστικού τομέα σε, τρίτους, σε τρίτες χώρες. Δεύτερον, θα καταθέσει μια τροπολογία σχετικά με τη συμμετοχή ε, των γυναικών ε, στις ε, ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Κάθε διαπραγμάτευση όπου εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην συμμετοχή των γυναικών ως παράγοντα επιτυχίας ε, για μια ειρήνη ε, που θα διαρκέσει και να υπάρξει μια καλή μετάβαση προς αυτήν. Τρίτον, θα πρέπει να περιλάβουμε την κατάσταση των ε, προσφύγων γυναικών και ετούντων εσύλο ε, και τα κράτη-μέλη ε, και ε, οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό και να λάβουν την επαρκή κατάρτιση για να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση των γυναικών. Και τέλος θα προσθέσει, μία παράγραφο σχετικά με την καταπολέμηση του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων καθώς επίσης ε, και μία παράγραφο σχετικά με τους ε, εξαναγκαστικούς ε, γάμους. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ε, έχω την ε, χαρά που είμαι σκιώδης ε, σε αυτή την έκθεση και θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερα θετικό το ότι επικεντρωνόμαστε στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία καθώς επίσης στο ζήτημα της, σεξου, της σεξουαλικής βίας ως ε, όπλο πολέμου. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν, όπως επίσης και η κατάσταση των ε, γυναικών προσφύγων, νεαρών κοριτσιών προσφύγων, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν ε, τα κορίτσια Ρωμά, καθώς επίσης και το τράφικινγκ, η πορνεία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και την απειλή από την ακραία δεξιά και το πόσο ε, οι ομιλίες μίσους τους επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των γυναικών προσφύγων ε, καθώς επίσης και για την κατάσταση των γυναικών σε κατεχόμενες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το κείμενο αυτό είναι ήδη αρκετά καλό. Ε, βέβαια θα το βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ με όλες μας τις ε, συνεισφορές. Έχω συνηθίσει τη συνεργασία με την Μπέατρης, οπότε αυτό διευκολύνει κατά πολύ το έργο μας. Έχουμε οπτική, όμοια οπτική γωνία για αρκετά ζητήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες πρόσφυγες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμπεριλάβουμε στις τροπολογίες μας. Ε, τις οποίες ε, θα ε, υποβάλουμε μεθαύριο. Επίσης, πέρα των όσων έχουν αναφερθεί ήδη, θα ήθελα να προσθέσω επίσης να υπάρχει μία αναφορά για την εκπαίδευση ενηλίκων, ιδιαίτερως για τις γυναίκες, αλλά και για τα παιδιά σε νοσοκομιακή εκπαίδευση ε, για παράδειγμα ε, ο νοσοκόμος δάσκαλος ε, είναι μια εικόνα που δεν έχουμε ιδιαίτερα συνηθίσει στην Ευρώπη όμως θα πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο καθότι φτάνουν πάρα πολλές γυναίκες στην Ευρώπη Επίσης όσον αφορά τις ανάγκες τους ε, και αυτό θα πρέπει να ε, περιληφθεί ενώ επίσης θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση στην κοινοβουλευτική διπλωματία όταν έχουμε να κάνουμε αυτά τα ζητήματα καθώς επίσης και ε, όλες τις ανησυχίες που σχετίζονται με τις ανησυχίες της ομάδας μου. Πέραν τούτου, έχουμε κάποιες τροπολογίες που είναι όμοιες με αυτές που ανέφερε η κυρία Μπιόρκ. Ε, αντιμετωπίζουμε ε, κάποια πράγματα με την ίδια λογική, όμως θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όμως θέλουμε να υπάρχει αναφορά ε, στο κείμενο και για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ενημερωτικά να σας πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 13 Οκτώβρη, 5 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπεφέρα έχει κάποια παρατηρήση μετά από αυτά που ακούσαμε. Βλέπουμε το κεφάλι όχι, οπότε τελειώσαμε αυτό το σημείο της ημερήθειας διάταξης και θα ξαναρχίσουμε αύριο το πρωί στις 10. Ευχαριστώ πολύ για... Όχι, διορθώνει η πρόεδρος στις 9. 10 θα ήθελα εγώ, λέει η πρόεδρος. 9 ώρα λοιπόν το πρωί Σας ευχαριστώ.